Good morning, ladies and gentlemen. Can Εγκρίνουμε την μίση διάταξη, σας παρακαλώ, γρήγορα, γρήγορα. Δεν έχω καμία καινούργια ανακοίνωση, υπάρχει αναμετάδοση στο κτλ. Πρώτο θέμα, ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για τη στρατηγική για την ενιαία αγορά. Ο εισηγητής Λάρκο. E Ευχαριστώ, ε, καλημέρα σε όλους. Όντως σήμερα ξεκινάμε τη νέα δική μας κοινοβουλευτική διαδικασία με αυτήν την ανταλλαγή απόψεων που για μας ε, σίγουρα είναι πολύ σημαντική. Ήδη είχα μία ε, συνάντηση με την Επίτροπο Μπιανκόφσκα αυτό το θέμα που μετά ήρθε να παρουσιάσει αυτή την στρατηγική στην Επιτροπή. Ξεκινώ με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και μετά θα μπω στην ουσία. Καταρχήν 25 Ιανουαρίου θα υποβάλω το σχέδιο έκθεσης στην Επιτροπή. Στις 27 του Ιανουαρίου έχουμε διοργανωμένη ακρόαση που, από το ΕΛΚ. Τέλη Φεβρουαρίου άλλη μια ακρόαση που διοργανώνει η Επιτροπή ΙΜΚΟ και στι 25 Φεβρουαρίου έχουμε την προθεσμία για υποβολή τροπολογιών. Μάρτιο-Απρίλιο θα εξαλλογήσουμε τις τροπολογίε και τις συμβιβαστικέ για να φτάσουμε στην υιοθέτηση στην Επιτροπή στι 21 Απριλίου για να περάσει από την Ολομέλεια τον Μάιο. Είναι αρκετά στενό αυτό το χρονοδιάγραμμα και γι' αυτό χρήσιμο είναι σήμερα να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μα για την ανταλλαγή απόψεων. Να μπω στην ουσία. Η ολοκλήρωση της ε, εσωτερικής αγοράς ήταν ανέκαθεν ένα σημείο κλειδί για αυτή την Επιτροπή και η Επιτροπή Γιούνκερ ε, θέσε σε εφαρμογή σημαντικές δράσεις που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει όλα ένα και περισσότερο να εκτελούνται. Στόχος είναι να βρεθούν μέτρα μέσω της καινοτομίας που να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα της μικρομεσαίας τις οποίες έχουμε προσέξει πολύ, δημιουργία νέων οικονομικών οντοτήτων που θα μπορούσαν να είναι οι startup, σε, αυτές, ε, σε αυτές ε, αφιερώνει ad hoc κονδύλια η Κομισιόν ακριβώς επειδή αυτές αντιπροσωπεύουν τον βιομηχανικό μας ιστό και έχουν και στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης κυρίως τη στιγμή που είναι νεανική ανεργία ε, φτάνει σε τέτοια επίπεδα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένα τι πρέπει να κάνουμε για τις μικρομεσαίες και τις καινοτόμες να εταιρείε, γιατί διαφορετικά μπορεί να δημιουργήσουμε σύγχυση χωρίς να έχουμε αποτελέσματα. Πρώτον, διαφορετικά εθνικά φορολογικά καθεστώτα. Αυτό είναι όντω ένα εμπόδιο στην εσωτερική μας αγορά. Οι επιχειρήσεις ε, ε, προσκρούν σε πολλά προβλήματα εάν θέλουν να μετακινηθούν από το ένα στο άλλο και έχουμε λοιπόν εμείς το καθήκον και την υποχρέωση να προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε τα φορολογικά καθεστώτα. Γνωρίζω πολύ καλά ότι εφόσον δεν υπάρχει πολιτική ένωση και δεν υπάρχει και φορολογική ένωση, αυτό καθίσταται περίπλοκο. Ένα πρώτο βήμα είναι να ε, φτιάξουμε έναν ενιαίο φόρο στο e-commerce, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ως μια πιλωτική δράση ε, μέσα σε άλλα θέματα που δεν θα μπορούσαν να είναι αρμοδιότητα της ε, ΙΜΚΟ. Να χρησιμοποιήσουμε επίσης ε, από πλευράς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τα ευρωπαϊκά κονδύλια να απλοποιηθούν, να είναι πιο προσιτά στους μεμονωμένους επιχειρηματίες. Για τις startup και τις μικρομεσαίες πρέπει να συντονιστούν καλύτερα και να δημιουργεί, δηλαδή, δημιουργηθεί ένα σύστημα επικοινωνίας μεταξύ τους, γιατί αλλιώς ο καθένας τραβά το δρόμο του. Αυτό αναφέρεται σε καλύτερη ρύθμιση και καλύτερη ρυθμίσει και απλοποίηση που είναι κλειδί για την δική μα θητεία, γιατί συχνά ψηφίζουμε χρήσιμε οδηγίε που όμω δεν εφαρμόζονται, όπω αυτή για τι κρατικέ προμήθειε, αλλά και ένα σωρό άλλε. Ένα σημαντικό θέμα που είναι και δικό μου προσωπικό πρόβλημα είναι ε, διαρκώς η καθυστέρηση ε, των πληρωμών. Δεν είναι δυνατόν να, να ε, πτωχεύουν εταιρείε λόγω των πιστώσεων και όχι των χρεώσεων. Το κράτος ζητά τους φόρους γρήγορα και άμεσα από την κάθε επιχείρηση, αλλά εν τω μεταξύ δεν πληρώνει το ίδιο και και στο υποχρεώσεις. Ε, καλύτερη διαχείριση λοιπόν με ένα μέσο το οποίο μπορούμε να εισάγουμε. Για την οδηγία για τις υπηρεσίες που είναι εξαιρετικά σημαντική είναι μια οδηγία που εφόσον δεν υπάρχει εναρμόνιση του συστήματος των υπηρεσιών στα μέλη να αντιμετώπισε προβλήματα. Πάντοτε λοιπόν στην κατεύθυνση της βοήθειας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει και για αυτήν να το σκεφτούμε και να αναλύσουμε πού λειτουργήσε και πού όχι. Σημαντικό και συμφωνώ με την Επίτροπο είναι το διαβατήριο υπηρεσιών, service passport, δηλαδή οι ίδιοι κανόνες και η ίδια εγγράφα για όλους όταν θέλουν να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση σε ένα κράτος μέλος. Να αφήσουμε και την συνεργατική οικονομία που είναι σημαντική ε, και δίνει συμβάλλει στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Ωστόσο, πρέπει να βρούμε στοιχεία των, των, τομέων κλειδιών, γιατί διαφορετικά φτιάχνουμε ακόμα περισσότερη σύγχυση, πράγμα που δεν εξυπηρετεί κανέναν. Τις προδιαγραφές ε, εγώ το έχω παρακολουθήσει από την προηγούμενη ε, θητεία, είναι σημειοκλειδί, βρισκόμαστε σε μια αγορά, πρέπει να έχουμε και ενιαίες προδιαγραφές και στις διαπραγματεύσεις για το TTIP και ζητάμε από τις ΕΠΑ να, να ομοιογενοποιήσουν τις προδιαγραφές τους, αλλά εμείς εδώ δεν το κάνουμε. Θα πρέπει λοιπόν να το στηρίξουμε αυτό και να καταστήσουμε πιο οικονομικό το σύστημα αυτό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, εποπτεία της αγοράς, το έχουμε πει επαναλημμένως, ιδιαίτερα μετά την υπόθεση Volkswagen, πρέπει να κλείσει αυτό το ευλογημένο ντοσιέ, το οποίο έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο εδώ και χρόνια και πρέπει να λύσουμε και το θέμα του άρθρου 7 στο εσωτερικό της ε, εποπτείας αγοράς και να μπλοκάρει αυτό ολόκληρο το φάκελο ε, το θέμα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ησυχάσουν γιατί από αυτό το κοινοβούλιο ε, επανειλημμένως είχε ψηφίσει για το Made in. Ναι, τώρα, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Ε, σας μίλησα έτσι γρήγορα, αλλά θέλω την άποψή σας για όλα αυτά. Ε, τώρα, οι διακρίσει ει βέρο των καταναλωτών είναι επίση σημαντικό. Έχουμε διαφορετικέ τιμέ και κόστη εργασία, γραφειοκρατία και όλων ε, των πάντων στα κράτη-μέλη και αυτό ε, καθιστά, δημιουργεί μάλλον ανταγωνισμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη, ενώ αντίθετα θα έπρεπε ο ανταγωνισμό να είναι ανάμεσα στι υπήρου. Αυτό πρέπει να πετύχουμε ε, και να ε, καταστεί πιο αποτελεσματική αξιολόγηση του geo-blocking, όπως ναι, λέγεται. Δεν θέλω να παρατείνω αυτές τις εξηγήσεις, γιατί και οι συνάδελφοι Σκιώδης έχουν το έγγραφο της Κομισιόν και με θα ήθελα να ακούσω την γνώμη τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Μάλιν Μίτσι. Ευχαριστώ. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις διότι αφορά όλες τις επιχειρήσεις και αυτές αφορούν όλους τους καταναλωτάς και καταναλωτρίας. Η σωστή λειτουργία της ενιαίας αγοράς εξαρτάται από την ανταπόκριση που θα έχουμε στις προκλήσεις του μέλλοντος. Γι' αυτό χαιρετίζουμε αυτή την πρόταση της Καμισιόν αλλά η πρόοδος αυτή δεν πρέπει να θεωρηθεί δεδομένη διότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά τις επιχειρήσεις και μειώνει την ανάπτυξη και άρα βλάπτει τους πολίτες. Σε πολλές χώρες δυστυχώς υπάρχουν λαϊκιστέ και λαϊκίστριες και οι οποίοι αντιτίθενται στην ενιαία αγορά και τα επιτεύγματά της. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Και δεν μπορούν οι χώρες μέλη επίσης να αντιμετωπίσουν τις μεταναστευτικές πλέον ροές και τους πρόσφυγες. Όλα αυτά δημιουργούν μια επικίνδυνη κατάσταση στην Ευρώπη που θα μπορούσε να οδηγήσει στη διάλυση όχι όμως της ενιαίας αγοράς αλλά και της ένωσης της ίδιας. Η έννοια αγορά θα μπορούσε όμως να είναι ένας από τους κύριους καταλήτες για την οικονομική αναθέρμανση και ανάκαμψη. Και γι' αυτό χαιρετίζω το γεγονός ότι η Καμισιόν μιλάει συγκεκριμένα για βαθύτερη ενιαία αγορά, βαθύτερη και δικαιότερη. Πρέπει όμως να εκφράσω και κάποια απογοήτευση γιατί δεν υπάρχει πολύ μεγάλη πολιτική θέληση για να τα πετύχουμε όλα αυτά. Αυτό πρέπει να το πρασέξουμε. Συνδέει η Κομισιόν μόνο με την οικονομία την ενιαία αγορά. Χρειάζεται η ενιαία αγορά βέβαια, όχι μόνο ανάπτυξη, αλλά και δημιουργία θέσεων απασχόλησης προστασία των καταναλωτριών και προστασία του περιβάλλοντος. Χρειάζεται η σωστή εξοικονόμηση μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Βαθύτερη και δικαιότερη ενιαία αγορά λοιπόν για μια στεναρότερη ευρωπαϊκή οικονομία με δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης και ευκαιριών καθώς και γενικώ καλύτερη διαβίωση για τους πολίτες. Δυστυχώς όλα αυτά δεν την χάνουν και σωστής εφαρμογής, διότι τα κράτη-μέλη δεν μεταφέρουν και δεν εφαρμόζουν όλα τα νομοθετήματα για την ίδια αγορά, δεν υπάρχει εναρμόνιση μεταξύ χωρών μελών και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημίες. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το αποφύγουμε στην πράξη έχουμε τα εργαλεία για να διασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, αλλά στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί πολύ καλά η ενιαία αγορά για μένα. Πολλοί φραγμοί δεν μπορούν να αρθούν παρά μόνο με την πλήρη εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας και του ισχύοντος νόμου για τον ανταγωνισμό. Παραδείγμα της χάρη. Όταν μιλάμε για το geoblocking, Πρέπει να σας πω ότι οι αθέμητες πρακτικές, η οδηγία για τους καταναλωτές λοιπά υπάρχουν, αλλά δεν δίνεται η κατάλληλη βοήθεια στα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να εφαρμόσουν σωστά αυτά τα νομοθετήματα. Αναμένω περισσότερο από την Καμισιόν για να μπορέσουμε να έχουμε θετικές επιπτώσεις από την λειτουργία της ενιαία αγοράς και τη ζωτή εφαρμογή της στρατηγικής του 2020 χρειαζόμαστε συγκεκριμένες προτάσεις με συστηματική έμφαση σε καλύτερη εφαρμογή των ισχυρών των κανόνων και με πιο στενά χρονοδιαγράμματα αυστηρά. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, Ευχαριστώ, Ντάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλο επιτεύγμα αυτή η ενιαία αγορά. Έχουμε προχωρήσει πολύ. Αλλά δεν αρκεί κιόλα. Εγώ σε σχέση με την ενιαία αγορά πιο πολύ σκέφτομαι τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις, γιατί οι μεγάλες έχουν περιθώριο να διακινήσουν όπως το εννοούν την, τα εμπορεύματά τους. Και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να εστιαζόμαστε πως πράττει και τη συγχαίρω γι' αυτό η συγκέντρια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα θα πρέπει να δούμε λοιπόν την δυνατότητα για παροχή καλύτερης υπηρεσίας και προς τις ε, μικρές επιχειρήσεις που μπορούν έτσι να μεγαλώσουν αλλά και προς την, ε, τον καταναλωτή. Δεν πρέπει να επιβαρύνεται βέβαια ο φορολογούμενος ε, από οποιαδήποτε υποστήριξη θα προσφερθεί, γιατί αρκετά δυσκολεύεται ήδη, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και την ε, υιοθέτηση της πρότασης για το SUP στην εποχή του ίντερνετ δεν είναι δυνατόν να χρειάζεται ε, να περάσει κανείς από τόσο διαφορετικές διαδικασίες για να καταγραφεί. Ε, στις νεοφυείς επιχειρήσεις είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον να υπάρξει υποστήριξη. Στις μεταφορές υπάρχει μεγάλο πεδίο για ε, βελτίωση. Πρέπει να δούμε πού εστιάζεται περισσότερο η ε, ζήτηση. Στη συνεργατική οικονομία θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι εάν νομοθετήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο Υπάρχει κίνδυνος να υπονομεύσουμε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσομένους τομείς της ευρωπαϊκής ε, οικονομίας. Πολύ προσεκτικά λοιπόν θα πρέπει να διαχειριστούμε τα θέματα αυτά και τα νομικά προβλήματα ασφαλώς έχουν ε, χαρακτήρα και πολύ τοπικό και θα πρέπει και αυτό να το δούμε. Στην υλοποίηση, συμφωνώ με τα σχόλια της ε, εισηγητρίας, εάν δεν υλοποιεί την νομοθεσία, ποιος ο λόγος να την εγκρίνουμε. Και βέβαια πρέπει να συνεργαστούμε επικοδομητικά με τα κράτη-μέλη ώστε να καλύψουμε τα θέματα των ε, ε, παραβιάσεων της εσωτερικής αγοράς χωρίς να χρειάζεται να προσφεύγουμε στα δικαστήρια. Καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ένα γνήσιο πρόβλημα και σοβαρό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα θεσμικά όργανα άλλωστε έχουν ε, πολύ κακές επιδόσεις, καθυστερούν δηλαδή ιδιαίτερα στις πληρωμές τους προς τους ε, ε, μικρότερους εργολάβους. Πρέπει λοιπόν και αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Η εσωτερική αγορά χρειάζεται να προχωρήσει, να προσελκύσει επενδυτές και για αυτό το λόγο κάποιες προτάσεις υπερβολικής εναρμόνισης στο ηλεκτρονικό εμπόριο με ανησυχούν γιατί κινδυνεύουν να σχηματίσουν φραγμούς και εμπόδια στην ε, ε, λειτουργία των επιχειρήσεων. Εν πάση περιπτώσει όμως υπάρχει ένα περιθώριο, κοιτάξουμε μόνο το ηλεκτρονικό εμπόριο και τον κίνδυνο για την επιβολή διακρίσεως εις βάρος ε, των παρόχων αντίστοιχων υπηρεσιών λόγω με το αν παρέχονται υπηρεσίες διαδικτυακά, διαγραμμικά ή μη, ε, πρέπει να προσέξουμε. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες ταυτόχρονα δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο και εκτός. Η Facebook και η Google, παραδείγματι, μπορεί να θεωρούμε ότι είναι μόνο διαγραμμικές, ε, έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την παραδοσιακή και μη διαγραμμική εμπορική υπηρεσία μέσω των διαφημίσεων αναπτύξει. Εν πάση περιπτώσει, οι προτάσει τη Επιτροπή εν μου φαίνονται ευπρόσδεκτε. Πρέπει όμω να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί δεν θα πρέπει να υπονομεύσουμε υφιστάμενα ε, εμπορικά και επιχειρησιακά μοντέλα. Βέβαια, η κινητικότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την εισηγήτρια. Περιμένω τις ε, απαντήσεις της φυσικά και ιδιαίτερα θεωρώ καλή ευκαιρία τη σημερινή συζήτηση. So for the GUE group it's Ines Suba. GUE, Suba. Not here. Ναι, είναι εδώ. Άλντε. Antonis No. Okay. Δεν είναι κανείς από την Άλντε. Ρίδα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή. Προσδοκώ δε το σχέδιο έκθεσής του. Η στρατηγική για την ενιαία, στη στρατηγική για την ενιαία αγορά χαιρετίζουμε το στόχο να είναι βαθύτερη και δικαιότερη γιατί είναι σημαντικό αυτό για την αποδοχή της από τους καταναλωτές και τις καταναλώτριες αλλά και το λαό γενικότερα για να μην έχουν την εντύπωση ότι μόνο οι επιχειρήσεις και τα κεφάλαια κινούνται ελεύθερα αλλά και οι άνθρωποι και οι άνθρωποι οι ίδιοι. Η άνηση μεταχείριση με βάση την εθνικότητα και την παραμονή, την εγκατάσταση είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και το geo βέβαια, αλλά όχι μόνο. Βέβαια από την άλλη μεριά υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουν γεωμπλοκαριστεί επιχειρήσεις γιατί ίσως δεν υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα, ας πούμε μια μικρή εταιρεία δεν μπορεί να συμμορφωθεί με το καθεστώς ΦΠΑ και αυτό αποφασίζει να μην πωλήσει σε κάποιες χώρες αλλά υπάρχει και geoblocking απλώς γιατί μια επιχείρηση μπορεί να προσπαθεί να κατακαιρματίσει την αγορά. Αυτό είναι αθέμητο, αθέμητο. Εμείς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και τη συμμόρφωση και την νομοθεσία. Επίσης η δέσμη για την κυκλική οικονομία έχει επιστρέψει και αυτό είναι καλό, αλλά η παλαιότερη πρόταση που αποσύρθηκε για την κυκλική οικονομία μας έδωσε την εντύπωση από τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο Τίμερμανς ότι θα ερχόταν στη συνέχεια ένα πιο φιλόδοξο πρόγραμμα και αυτό δεν το βλέπουμε. Και εδώ πρέπει να τα πει αυτά το κοινοβούλιο για την sharing economy πρέπει να διαφοροποιηθούμε, να διαφοροποιήσουμε τις προτάσεις μετά από τις ε, διαβουλεύσεις και για την ενιαία ψοφιακή αγορά. Ο, να πούμε ότι δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις και πλατφόρμες το ίδιο. Μπορεί να έχει ιδιαίτερα δικά της προβλήματα η sharing economy και στις προκλήσεις προς τον ανταγωνισμό. Παραδείγματο χάρη να μιλάμε για την διαλειτουργικότητα interoperability να έχουν πιο εύκολα τη δυνατότητα οι επιχειρήσεις να περάσουν από τον ένα ανταγωνιστή στον άλλον ή οι καταναλωτές μάλλον και επίσης πρέπει να δούμε τι συμβαίνει με τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε χωριστούς τομείς, χωριστά. Όσο για τις βέλτιστες πρακτικές, η διευκόλυνση των δημοσίων προμηθειών και της εποπτείας της αγοράς είναι γνωστή, αλλά έχουμε μερικές ανησυχίες ως προς το πώς θα γίνει ακριβώς η εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής βασικά η αρχή follow the money είναι σωστή. Δεν σημαίνει βέβαια ότι θα παρακολουθούμε μέχρι και την κραβατοκάμαρα τη συμπεριφορά των καταναλωτριών, αλλά είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η παραχάραξη και η παραβίαση και η απάτη δεν είναι ακριβώς το ίδιο μεταξύ τους. Ας πούμε τα γενώσιμα φάρμακα. Μία παραβίαση σε μία χώρα δεν παραπλάνει αναγκαστικά τον καταναλωτή αν γνωρίζει τι ακριβώς παραχάραξη έγινε. Βεβαίως, για τους ενδιάμεσους δεν πρέπει καμία επιχείρηση να μπορεί να παίξει το ρόλο του δικαστηρίου. Το Κοινοβούλιο απέριψε πριν από μερικά χρόνια την ιδέα του patented software, του λογισμικού με πνευματικά δικαιώματα. Αλλά αποσιοποιητικά. Επίσης η Κομισιόν μίλησε για την αναθεώρηση της, ναι. της διαδικασίας για το διαβατήριο υπηρεσιών. Εμείς είμαστε υπέρ της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών, αλλά πρέπει οι κανόνες να τηρούνται και στη χώρα προορισμού και όχι μόνο προέλευσης όπως λέει η οδηγία για τις υπηρεσίες. Ας μην το ξανανοίξουμε όμως αυτό τώρα. Επίσης για την αμοιβαία αναγνώριση Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η αρχή της εποπτείας των αγορών θα κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει και θα ελέγχει πράγματι τη συμμόρφωση των προϊόντων ως προς τα πρότυπα. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της ομάδας μου και πιστεύουμε ότι μπορούμε τελικά να καταλήξουμε σε μία δέσμη που όντως να εμβαθαίνει και να καταλήγει σε δικαιότερη ενιαία αγορά. Ευχαριστώ, Τζούλια. Επόμενο, ε, στη, στη λίστα των σκεδών είναι ο Μάρκο Ζουλό. Και μετά η ε, Μαλίν Τροσκέντσκι. Όχι, δεν είστε εδώ. Θέλει κάποιος άλλος. Η Άννα Μαρία Κοράτσαμπελ. Θα σας διαβάσω τον κατάλογο. Κοράτσαμπελ, Σενφίλτ, Σαλτομόσα, Γιακονσάρι, Ντάντι. Okay. Άννα Μάρια Ευχαριστώ πολύ. Εγώ συμφωνώ με το όσα είπαν οι συνάδελφοι. Καλωσορίζω και στηρίζω αυτή τη στρατηγική που προτείνει η Κομισιόν για την αναζωγόνηση της ενιαίας αγοράς. Τα όσα λέει, πολλά μάλλον από αυτά που λέει η Κομισιόν, η Επιτροπή μας έχουν συμπεριληφθεί και αυτό είναι πολύ θετικά, αλλά μας ε, μας ε, κάνει να μπορούμε τόσο λίγα συμβαίνουν. Ελπίζουμε πως αυτή η στρατηγική θα βοηθήσει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε κομισιόν και κοινοβούλιο και να ζητήσουμε λογαριασμό από τα κράτη-μέλη για το κόστος της μη Ευρώπης βασικά. Εάν δεν σοβαρέψουν τώρα όπου τα χρήματα των φορολογουμένων είναι πια λιγοστά και δεν έχουμε ακόμα βγει τελείω από την κρίση και πρέπει να δώσουμε δουλειές στους πολίτες μας αλλά και στους πρόσφυγες που καλωσορίζουμε στην Ευρώπη αν δεν χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό της, ε, της ενιαίας αγοράς έρωτας τους φραγμούς, τα εμπόδια που την επηρεάζουν την ενιαία αγορά δεν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε νομίζω. Γενικό μου σχόλιο είναι λοιπόν ότι συμφωνώ με την πρόταση της Κομισιόν αλλά ότι εγώ θα ήμουν ακόμα πιο ε, ριζοσπαστική γιατί τα λέμε αυτά εδώ και χρόνια και δεν νομίζω πως αρκούν. Ε, καλωσορίζω την εστιασμό στην επιβολή, καλύτερη εφαρμογή, καλύτερη εκτέλεση, ε, ε επίσης ε, έμφαση στις υπηρεσίες, στην εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, ιδιαίτερα η πρόταση για αύξηση και διεύρυνση της διαδικασίας κοινοποίησης στην, στην οδηγία για τις υπηρεσίες, δυνατότητα μεταφοράς και γεωγραφικό μπλοκάρισμα, πολύ σημαντικό. Επίσης, η πολιτική μηδενική ανοχής, γιατί η Κομισιόν είπε ότι πρέπει να αλλάξει νοοτροπία στα κατημέλη. Δεν είναι θέμα ανάλυσης, όχι. Είναι θέμα έναρξης ε, διαδικασιών κατά παράβαση και εφαρμογής αυτών. πραγματικά καλωσορίζω το γεγονός ότι ο τομέας λιανικής πώλησης για πρώτη φορά έχει συμπεριληφθεί σε μια στρατηγική της ε, Κομισιόν για την ενιαία αγορά και νομίζω ότι εμείς εδώ, χάρη σε εμά έγινε μάλλον αυτό, στη δική μας Επιτροπή, υποστηρίζω το κομμάτι αυτό γιατί το ηλιανικό εμπόριο, απλά ε, τα μέτρα για την ε, δημιουργία είναι κάπως αδύναμα ο αριθμός προστατευτισμού που έχουμε για τομέα της, της ε, για, τη δημιουργία και κατάσταση εταιρεία ε, είναι κάπως αδύναμος αυτός ο τομέας λοιπόν και θα πρέπει να το ξαναδούμε. Τώρα συμφωνώ για την ε, οικονομία την ψηφιακή. Ε, σωστό είναι να την παρακολουθούμε ε, ε, γιατί αναπτύσσεται, αλλά δεν πρέπει να την δέσουμε με νομοθεσία. Θα πρέπει πολύ καλά να το εξετάσουμε πριν κάνουμε πράγματα σε νομοθετικό επίπεδο στην, στην Ευρώπη. Τώρα, νέο εργαλείο για την αγορά ε, δεν ξέρω ακριβώ τι εννοούμε με όλα αυτά που λέμε εδώ. Πάντως αυτό που θέλω να πω είναι βεβαίως ε, το θέμα της ενιαίας αγοράς. Μιλάμε για το θέμα αυτό χωριστά βέβαια, αλλά είναι καλό που έχει μπει τώρα στην ανακοίνωση και η ελεύθερη μετακίνηση των ε, στοιχείων, των δεδομένων είναι το ίδιο σημαντική με όλες τις άλλες ελεύθερες μετακινήσεις στην εποχή μας. Τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την νέα αγορά γιατί εμπνέει την ε, προστασία των δεδομένων και είναι θέμα της ΛΥΜΠΕ. Αυτό διέπει ολόκληρη την ψηφιακή αγορά. Εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσφέρουμε νομική βεβαιότητα και γρήγορα. Ελπίζω πως θα εγκριθεί μέσω των τριμερών διαλόγων μέχρι τα τέλη του έτους. Με ασφαλή λιμένα. Και αυτό ε, ε, επηρεάζει κάθε μια επιχείρηση που εξάγει στην Ευρώπη. Υπάρχει ένα νομικό κενό λοιπόν εδώ και το έγγραφο της Κομισιόν στις 6 Νευρίου δεν αρκεί για να καλύψει την επίπτωση της απόφασης του δικαστηρίου στην ευρωπαϊκή οικονομία. Τελευταία μου παρατήρηση είναι ότι πρέπει να είμαστε καλύτεροι στο να ενημερώνουμε για τα ωφέλη της ενιαίας αγοράς και τα εργαλεία που έχουμε στη θέση μας, όπως το Solvit και άλλα ψηφιακά εργαλεία που είναι παντελώς άγνωστα στους πολίτες αλλά και στις εταιρείες. Ε, κάτι το, θέλω να ευχαριστήσω την Λάρα Κόμη για μια πολύ καλή αρχή γιατί ξεκίνησε την εργασία σε αυτό το θέμα στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ ευχαριστώ. Σένφιλντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει δυστυχώς να σημειώσω ότι οι χειμερινοί μήνες δεν ε, αποτελούν πηγή αισιοδοξία και μάλλον είναι καταθλιπτικοί. Όπως άλλωστε και το συγκεκριμένο έγγραφο. Δεν βλέπω να εκθέτει τίποτε διαφορετικό από τα τετριμένα για την αποτελεσματική λειτουργία της ιστορικής αγοράς. Για μένα ο ιός ο οποίος έχει πλήξει την εσωτερική αγορά είναι οι υπερβολικές ρυθμίσεις και ο υπερβολικός προστατευτισμός. Κάθε διάταξη και κάθε κανονισμός οδηγεί σε νέες διατάξεις και σε νέους κανονισμούς, όλο και πιο λεπτομερείς. που φτάνουν μέχρι του ε, ύφους των οδηγιών χρήσεως. Δεν είναι δίκαιο αυτό που παράγεται, οδηγίες χρήσεως είναι. Και αυτό προφανώς κάνει κακό και στις μικρές και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Έχουμε και τους εθνικούς προστατευτισμούς προστατευτισμό για τον οποίο φέρουν την ευθύνη όλα τα κρατη αν και ορισμένα είναι πιο ε, επιτυχή από άλλα. Και είναι προστατευτισμό σε δύο επίπεδα. Σε επίπεδο τύπου και σε επίπεδο ουσίας. Με όλη αυτή την νομοθεσία που εμποδίζει, παραφράσει, ε, παρακολεί την δραστηριότητα ξένων επιχειρήσεων από το ένα κράτος στο άλλο, παρά το γεγονός ότι εν λόγω ξένες επιχειρήσεις προέρχονται από μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι λοιπόν ό,τι και να κάνουμε, αν δεν πούμε ότι καταπολεμούμε τις υπερβολικές ρυθμίσεις και αυτή την υπερπληθώρα του ευρωπαϊκού, ε, της ε, ευρωπαϊκής νομοθετικής παραγωγής, δεν θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια αποτελεσματική εσωτερική αγορά και μια παγκόσμια ανταγωνιστική οικονομία. Το ξανά είπα και την άλλη φορά. Είμαστε κοινότητα. Δεν μπορεί μόνο η Γερμανία και η Γαλλία ή μόνο η Πολωνία και η Λιθουανία να λαμβάνονται υπόψη. Μία κοινότητα, μία οικονομία συνολικά που πρέπει να καταστεί επαρκώς ανταγωνιστική σε σχέση με τις λοιπές κοινότητες όπως είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε ή οι χώρες της Άπο Ανατολής όπως το Μεξικό. Έτσι λοιπόν το να περιοριζόμαστε και να επιμένουμε στο να δίνουμε οδηγίε χρήσεω στου επιχειρηματίε, δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτε σε σχέση με του μεγάλου ανταγωνιστέ όπω η Κίνα. Στι υπηρεσίε, Φερρυπίν. Που και την τελευταία φορά είχα επισημάνει ότι δεν έχω καταλάβει το σκοπό εξυπηρετεί η πρόταση. Γιατί τι να κάνουμε τη συζήτηση για την ε, εσωτερική αγορά όταν χρειάζεται ένα είδος διαβατηρίου για τις επιχειρήσεις. Όσο υπάρχει αυτή η ανάγκη για διαβατήριο για τις επιχειρήσεις, δεν θα υπάρχει εσωτερική αγορά. Γιατί δεν θα μπορεί η επιχείρηση με έδρα σε ένα κράτο μέλο να αναπτύσσει δραστηριότητε και τι υπηρεσίε τη σε ένα άλλο. Όσο χρειαζόμαστε λοιπόν έγγραφα, πιστοποιητικά, διαβατήρια, όπω θέλετε πείτε τα, δεν θα γίνεται σωστά η δουλειά, δεν θα υπάρχει σωστή εσωτερική αγορά. Τώρα, αν κατάλαβα καλά, κάποιος είπε ότι αυτό το διαβατήριο στόχο έχει να πιστοποιεί ότι ισχύουν οι ίδιες διατάξεις και κανονισμοί στη χώρα προελεύσεως και στη χώρα υποδοχής. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Θα προσπαθήσουμε να πατάξουμε τον ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει. Ο ανταγωνισμός είναι ζωτική λειτουργία της οικονομίας. Πρέπει να είναι διαφορετικές συνθήκες. Και μετά να διαλέξει ο καταναλωτής τι είδους υπηρεσία ή αγαθό θέλει να αγοράσει. Γιατί δεν θα έχει σημασία από πού θα αγοράζει, από ποιον θα αγοράζει, αλλά τι θα αγοράζει και το γεγονό ότι θα έχει την ελεύθερη επιλογή. Αυτό θα έχει τη ζωτική σημασία. Άρα ούτε διαβατήρια, ούτε οδηγίε χρήσεω, ούτε άλλες διατάξεις θέλουμε. Υπερβολικές ρυθμίσεις λοιπόν και η υπερπληθώρα αυτών καταστρέφει την εσωτερική αγορά μαζί με τον προστατευτισμό. Και δεν θα εκθέσω τα προβλήματα του τυπικού, του, τύπης, του διαδικαστικού δηλαδή ε, προστατευτισμού, αλλά του άτυπου που είναι και πιο επικίνδυνος. Φερρυπίν και θα αναφέρω τη Γαλλία συγκεκριμένα, εάν υπάρχει προϋπόθεση, χώρα, ε, εταιρεία η οποία αγοράζει υπηρεσία από άλλες επιχειρήσεις, να φροντίζει στη χώρα προελεύσεως ο παροχός των υπηρεσιών να συμμορφούνται προς τις δημοσιονομικές προϋποθέσεις ή τις φορολογικές και αυτές ποια χώρα μπορεί να αναλάβει δέσμευση σε σχέση με την τήρηση των φορολογικών υποχρέσεων του αντισυμβαλουμένου της και κυρίως αν αυτός ο αντισυμβαλόμενος προέρχεται από άλλη χώρα. Αυτός λοιπόν είναι ο άτυπος προστατευτισμός, ο οποίος εξασφαλίζει πως μια, μια επιχείρηση προερχόμενη από άλλη χώρα δεν θα μπορεί να συνεργαστεί με την επιχείρηση που ανέφερα νωρίτερα. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό και πώς θα αμφισβητήσουμε αυτούς τους τόσο επιβλαβείς κανόνες και αρχές. Εδώ είναι τα σοβαρά προβλήματα λοιπόν. Η διατάξη περί ελάχιστου μισθού. Φερρυπίν. Εκεί όπου μπορεί να υπάρχει η συνέπεια σε σχέση με τη λειτουργία των μεταφορικών επιχειρήσεων που θα καλούνται δηλαδή να τηρήσουν διατάξεις άλλου κράτους. Πρέπει λοιπόν, πρέπει λοιπόν να ε, σταματήσουν όλες αυτές οι τάξεις. Καλώς λέει ο Πρόεδρος να τελειώνουμε όμως γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Σας ευχαριστώ. Και εγώ εκτιμώ αυτή την νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά και συμφωνώ ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία αλλά και κάποια λιγότερο θετικά. Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Πήρα όμως το λόγο επειδή θέλω να εκφράσω την υποστήριξή μου προς την εισηγήτρια τη Λάρα Κόμη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να στείλουμε ένα μήνυμα και να πούμε πως επιτέλους κάτι πρέπει να κάνουμε ώστε η ενιαία χώρα να μπορέσει να λειτουργήσει και να υλοποιηθεί. Με όλες τις ε, τα συμπληρώματα από πτήρια της αγοράς. Για παράδειγμα, η ενιαία αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει μέχρι ότου να ολοκληρωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο. Άρα λοιπόν πρέπει στην έκθεσή μας να υπογραμμίσουμε ότι σήμερα, τώρα μάλλον πρέπει να κλείσουμε όλα σε αυτές τις ελλείψεις. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να εγκριθούν και να εφαρμοστούν νέοι κανόνες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Η στρατηγική είναι πολύ σημαντική. Θα δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση εάν και μόνο εάν εφαρμοστούν στην πράξη οι προτάσεις που διατυπώνονται εδώ. Παραδείγματος χάρη, ο κανονισμός για το ΦΠΑ πώς και πότε θα αλλάξει. Πότε και πότε. Γιατί είναι σημαντικό να γίνει εκεί μια μεταρρύθμιση. Η συγητής αναφέρθηκε στην καινοτομία. Η συγήτρια μάλλον η οποία συνίσταται στην shared economy. Στη Φιλανδία άκουσα άλλον όρο, jobbing economy, δηλαδή ότι θα αλλάξει και η αγορά εργασίας και οι σχέσεις εργοδοτών εργοζομένων. Θα δημιουργήσουν, λέει, και νέες δυνατότητες για μετανάστες, αλλά πώς πώς ακριβώς θα διευθετηθεί αυτή η νέα οικονομία. Υπερβολικά πολλή νομοθεσία μπορεί να την σκοτώσει, υπερβολικά λίγη να δημιουργήσει μια ζούγκλα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τη σωστή εξισορρόπηση. Και εδώ πρόκειται για τα πρώτα βήματα. Ευχαριστώ λοιπόν την Καμισιόν για τη στρατηγική που διατύπωσε. Πιστεύω ότι πρέπει τώρα οι προτάσεις αυτές κάποτε να εφαρμοστούν. Η Κλαντάντε. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να είμαι σύντομος. Είναι η έκθεση, νομίζω, μία έκθεση με πολλά φωτεινά σημεία και με πολλές σκιές ταυτόχρονα. Είναι καλό να είμαστε φιλόδοξοι όσο και επικίνδυνο. Πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθήσουμε να υψώσουμε λίγο τον πύχη των ε, αποφάσεών μας και γι' αυτό πιστεύω ότι η Επιτροπή μας ε, με την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές μπορούν να κάνουν μια σημαντική δουλειά με ένα σημαντικό και σαφές μήνυμα που μπορούμε να αποστείλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε χρονική στιγμή όπως η παρούσα και νομίζω ότι είμαστε λίγο φιλόδοξοι σε σχέση με την εσωτερική αγορά για τα αγαθά και την ανταγωνιστικότητα της παραγωγής της Ευρωπαϊκής. Η εσωτερική αγορά πιστεύω θα πρέπει να εξυπηρετήσει την ανάκαμψη της Ευρώπης και της ε, παραγωγής της, της Ευρώπης ως τόπου παραγωγής αγαθών ποιοτικών όπως και υπηρεσιών. Δεν μπορούμε να είμαστε δηλαδή μόνο μια εμπορική πλατφόρμα. Ένα όρεμα της Ευρώπης το οποίο θα πρέπει να εγγραφεί μέσα στην εσωτερική αγορά. Γιατί δεν είμαστε μόνο ένας χώρος ανταλλαγής των εμπορευμάτων που εμείς οι ίδιοι παράγουμε, η Ευρώπη. Πρέπει να δούμε και την ε, λειτουργία μας μέσα στην διεθνή αγορά και το διεθνές εμπόριο. Σε αυτό πρέπει να είμαστε κάπως πιο φιλόδοξοι και το είπε πολύ καλά, πολύ ευστοχά η συγγήτρια. Βλέπουμε από την έκθεση στοιχεία και ανησυχητικά αλλά και ε, θετικά. Έχουμε ένα 39% του ΑΕΠ που στηρίζεται σε διανοητική παραγωγή Έχουμε μεγάλο ποσοστό το οποίο, ε, ΑΕΠ που προκύπτει σε σχέση με προϊόντα παραποίησης ή καταστρατήγησης των διατάξεων και αντιγραφής της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας. Και εδώ θα πρέπει ιδιαίτερως να πιέσουμε για την οδηγία για την εποπτεία των αγορών, συμπεριλαμβανομένου και το άρθρο 7 και αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι μάλλον διστακτικά βήματα και το λέω ευγενικά σε σχέση με αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενώ έχουμε τοποθετηθεί πρόσφατα, πριν από μερικούς μήνες, με πολύ με συντριπτική πλειοψηφία σε σχέση με τους καρόνες προέλευσης για τα μη γεωργικά προϊόντα, ήταν σαφής τοποθέτηση του Κοινοβουλίου στην Ολομέλεια. Παρόλα αυτά λοιπόν βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για περαιτέρω μελέτες, αξιολόγηση κτλ. Τη βλέπουμε μάλλον διστακτική λοιπόν και δειλή στο, σημείο αυτό. Σε άλλα σημεία που μπορώ να κρίνω θετικά είναι η προσέγγιση του επαγγέλματος και εδώ θα υποστηρίξουμε και θα δώσουμε χείρα βοηθεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προχωρήσουμε και στον τομέα των επαγγελμάτων και της αναγνώρισης του σε μια εσωτερική αγορά και ένα τελευταίο σημείο για το sharing economy, που θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε και τη συζήτηση των τροπολογιών για την εσωτερική ψηφιακή αγορά τις τελευταίες ημέρες, όπου καλύπτεται σε έναν βαθμό και το θέμα αυτό και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια καλή συμβαστική λύση και μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει το θέμα αυτό να το προσεγγίσουμε με αποφασιστικότητα και με την ε, κατάληξη σε μια απελευθέρωση τέτοια που να μην στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, χωρίς ταυτόχρονα βέβαια να πέσουμε και στην παγίδα της περιβολικής ε, νομοθετικής ε, παρέμβασης. Χρειάζεται επομένω μια προσέγγιση που θα ενθαρρύνει αυτό το νέο τύπο οικονομίας χωρίς ταυτόχρονα να παρεμποδίζει την ανάδειξη και νέων δυνατοτήτων για τις υπηρεσίες. Πολλά έχουμε να κάνουμε ακόμα και ασφαλώς έχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις στα κράτη-μέλη. Αλλά θα ήθελα να σας αναφέρω ένα παράδειγμα δικό μου για τη διαχείριση λοιπόν επί 10 έτη των ε, αστικών συγκοινωνιών της Τοσκάνης έγινε μία προκήρυξη, ένας διαγωνισμός ε, πανευρωπαϊκός ε, με μία οδότη, μία γαλλική επιχείρηση, διαχείριση από το Παρίσι και, την, το μεγάλο Δήμο Παρισίων που ήδη έχει κτλ. Με εκχώρηση για 35 χρόνια χωρίς διαγωνισμό στη Γαλλία. Γιατί έτσι είναι η νομοθεσία. Εντάξει, λοιπόν, πρέπει να εξασφαλίσουμε έναν καλό ανταγωνισμό, έναν υγιή ανταγωνισμό, αλλά να αποτρέψουμε και τι στρεβλώσει του ανταγωνισμού και την κατάχρηση. Με μια υγιή αγορά. Όλα αυτά πρέπει να τα αξιολογήσουμε από κοινού και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει ε, θα χρειαστεί να, θέσουμε, να διατυπώσουμε περαιτέρω προτάσεις στη συνέχεια. Άντερσον. Εγώ πολύ καλωσορίζω αυτή την ανταλλαγή απόψεων για τη δουλειά που έχει κάνει η Συγήτρια και άλλοι για αυτό το θέμα. Πάντω είναι σίγουρο ότι η νέα αγορά είναι ένα από τα μεγαλύτερα μα εκπαιδεύματα, αλλά δεν είναι αυτό ο σκοπό, ωστόσο. Πρέπει να ε, κάνουμε μια αναδρομή σε τελευταία 15 χρόνια όσον αφορά στους αρχικούς στόχους της Λισαβόνας και συγκεκριμένα ότι θα πρέπει να έχουμε την πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία του κόσμου βασισμένη στη γνώση που θα μπορεί να δημιουργεί βιώσιμη ανάπτυξη, καλύτερες θέσεις απασχόλησης και καλύτερη κοινωνική συνοχή. Και πολλά από αυτά τα σημεία που αναφέρονται είναι χρήσιμα συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι ο κόσμος έχει το δικαίωμα ε, στην απασχόληση και αυτό το δικαίωμά του θα πρέπει να προστατεύεται σε ολόκληρη την Ένωση προς το συμφέρον της καλής διακυβέρνησης και του ισότιμου και αυτό ισχύει τόσο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και για όλες τις ε, επιχειρήσεις και καλωσορίζω την ε, αναφορά στο ότι θα πρέπει η ευρύνη αγορά να είναι πιο δίκη και αναφέρεται και στο κείμενο πρέπει να είμαστε ωστόσο ρεαλιστές για το που βρισκόμαστε. Ορισμένα τα προβλήματα οφείλονται στη δημοσιονομική κρίση, χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά δεν είμαστε και τα κρατημέλη άσχετα με όλα όσα συμβαίνουν και τη δημιουργία των ε, συνθήκων που μας έφτασαν εκεί. Θα πρέπει ωστόσο να αναγνωρίσουμε ότι 60 ε, εκατομμύρια κόσμος είναι άνεργος στην Ένωση ε, ότι θα πρέπει ε, να πάμε πίσω στις καλύτερες θέσεις απασχόλησης και τις περισσότερες. Πρέπει αυτό να είναι η έννοια. Όχι προστατευτισμός, αλλά η προστασία των καλών ε, συλλογικών συμβάσεων και των καλών ε, εργασιακών σχέσεων. Γιατί αυτό είναι η ουσία. Είμαστε λοιπόν σε, μια, θέματα τα οποία μας βρίσκουν σύμφωνος. Λάμπερτς Φαν Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να υπογραμμίσω την ε, δέσμευση, να υπογραμμίσω και να επενέσω την προσήλωση της ΛΑΡΑ σε αυτό το θέμα. Πρέπει να βρούμε ισορροπία ανάμεσα στην νομοθεσία και τη φιλοδοξία των επιχειρηματιών και κυρίως των νέων που ασχολούνται με τις διάφορες, που προβαίνουν μάλλον σε διάφορες πρωτοβουλίες. Θα πρέπει κανείς να καταρτιστεί για την νέα οικονομία που υπάρχει μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και στις υπηρεσίες, στην συνεργατική οικονομία. Θα πρέπει να γίνουν καινοτομίε. Χιλιάδες άνθρωποι ε, και νέοι μάλλον ασχολούνται με αυτά και έπειτα υπάρχει και το πακέτο πρωτοβουλίες για τις ε, startup. Τι κάνει ο κόσμος. Εγώ συμμετείχα σε μία συνάντηση στο, στη Λονδίνο ε, για τη startup και σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτοί, αυτές οι πρωτοβουλίες εξορισμού είναι διεθνείς γιατί οι νέοι και ο κόσμος στον οποίο ζουν είναι διεθνοποιημένος. Ε, και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Ο Κρούς έλεγε τότε ότι πρέπει να περάσουμε όχι μόνο από τη startup, αλλά να περάσουμε και για σε μια stand-up Europe, σε μια άλλου είδους Ευρώπη, γιατί η κλίμακα έχει αλλάξει. Θα πρέπει εμείς να προσφέρουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και ευρωπαϊκό κλίμακα. Εάν δεν το κάνουμε, ε, οι νέοι θα πάνε στις ΙΠΑ, όπου υπάρχουν αυτές, ε, αυτά τα φυτόρια, ε, οι επιχειρήσεις θα μεταφερθούν απλά στη Silicon Valley και θα ελπίζουμε μετά να επιστρέψουν. Αλλά είναι κρίμα, πολύ κρίμα. Το startup είναι πολύ σημαντικό και οι startup μάλλον είναι πολύ σημαντικέ και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τις στηρίξουμε οικονομικά, να προετοιμαστούμε για τα επόμενα 20-25 χρόνια όπου η βιομηχανία θα αλλάξει πραγματικά. Και υπάρχει εδώ μια δυνατότητα για όσους είναι πιο έτοιμοι πιο... και έχουν αυτή την αίσθηση της επιχειρηματικότητας. Πρέπει να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν, όχι μόνο στις Μητροπόλεις της Μεγάλες Πόλης, με τα διαρθρωτικά ταμεία, ας πούμε, μπορούμε να παρέμβουμε σε χώρες όπως η Ρουμανία, όπου υπάρχουν πρωτοβουλίες σε startup και φυτώρια. Και αυτό για να αποφύγουμε ικανοί νέοι να στερούνται μια βάση ενό ιστού, τον οποίο εμεί μπορούμε και πρέπει να οικοδομήσουμε. Και Λάρα, μπορείτε να βασίζεστε στη συνεργασία μου. Ευχαριστώ. Γιάννη Νίλσεν. Eh, Σα ευχαριστώ. Δεν είχα την πρόθεση να πάρω το λόγο, να ζητήσω το λόγο, αλλά ο Πολωνός συνάδελφος με όθησε να παρέμβω. Ελεύθερη αγορά κατεμένα δεν είναι κάτι που μπορεί να βιωθεί χωρίς κανόνες. Χρειάζεται διευθέτηση. Μία ελεύθερη αγορά χωρίς κανόνες καταλήγει να αυτοκαταστρέφεται. Χρειαζόμαστε λοιπόν διευθέτηση. Μιλήσατε για τις μεταφορές. Πράγματι υπάρχει ένα είδος κοινωνικό dumping στις μεταφορές σήμερα. Dumping. Έχω και εγώ γνωρίσει επιχειρήσεις και εργαζόμενους στον τομέα αυτών που μου λένε ότι ήδη υπάρχουν κανόνες. Αυτό που χρειάζεται είναι να εφαρμοστούν. Αυτό λείπει σήμερα. Και από την άλλη μεριά οι εργοδότες απίστευτο το ίδιο μου είπαν. Πρέπει δηλαδή να γνωρίζουμε σαφώς ποιοι κανόνες θα ισχύουν. Υπάρχουν επιχειρήσεις μεταφορικές σήμερα που λειτουργούν στη Σουηδία αλλά που βασίζονται, εδράζονται σε, ένα, σε μια ταχυδρομική θηρίδα στη Λιθουανία. Συμφωνώ ότι χρειάζεται καλύτερη διευθέτηση, πιο απλή κανόνες, πιο εύληπτη. Δεν χρειάζεται τεράστιος αριθμός καινούριων κανόνων, αρκεί να εφαρμοστούν οι ισχύοντες. Έπειτα η προστασία των καταναλωτριών. Και εδώ πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες είτε αγοράζει κανείς σε πραγματικό μαγαζί είτε από το ίντερνετ. Κοιτάξτε και εγώ θέλω να σας πω μερικά. Χωρίς να επαναλάβουμε τα εξαιρετικά επιχειρήματα που ακούσαμε ήδη. Θα ήταν χρήσιμο αν μιλούσαμε και για τις μη νομοθετικές πτυχές, γιατί είναι σημαντικές και αυτές ας πούμε στο 4.1 που γίνεται λόγος για συμμόρφωση. Αυτή τη συζήτηση την έχουμε ξανακάνει στην Επιτροπή μας για τις ελλείψεις των single points of contact. Η Κομισιόν μιλάει και για άλλα επίπεδα πληροφόρησης, να μας πει και γι' αυτό τίποτε παραπάνω. Και στο 4.2 μιλούν για γνωστοποίηση, notification, και εδώ θα ήθελα να καταλάβουμε μερικά παραπάνω πράγματα γι' αυτό γιατί θα μας βοηθούσε. Για το Service Passport τώρα έγινε λόγος ήδη για το ότι η χώρα προορισμού πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Πώς το Services Passport θα συνλειτουργήσει με τις επαγγελματικές κάρτες. Ιδίως για το θέμα home και host. Όσο για τον εξυγχρονισμό των προτύπων 3.1 Πρέπει να το αναλύσουμε χωριστά νομίζω. Τι εννοούμε ξεχρονισμό προτύπων. Ας πούμε για τις υπηρεσίες γίνεται λόγος για υπηρεσίες που βασίζονται στη ζήτηση. Ποιος όμως κάνει τη ζήτηση ο καταναλωτής ή ο προμηθευτής. Για την υποπτία της αγοράς συμφωνώ με την Αναμαρία. Δεν μπορούμε την έννοια του made in να την περιορίσουμε σε αυτά που προτείνονται. Πολλοί θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε και ότι η εποπτεία της αγοράς θα είναι πραγματική. Για τις δημόσιες προμήθειες το 3-2 νομίζω αν δεν απατιέμαι. Καλό θα ήταν να γίνει μια καλύτερη γνώση και για την προ, προεμπορικές προμήθειες. Υπάρχουν επίσης ορισμένα θέματα για την πρόσβαση στα patterns από τις μικρές επιχειρήσεις. Α, και αυτά ίσως θα έπρεπε να τα ξαναπούμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, να μας εξηγήσετε λίγο τι εννοείται και για τη διαδικασία refit. refit. Σας ευχαριστώ κύριε εισηγήτρια. Και τώρα η Κέρστεν Τζόνα από την Κομισιόν. Θα μιλήσει ή ο σύντροφός της εκεί. Α, ο σύντροφος, λοιπόν, κύριος Καμίνσκι. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια που περιέγραψε την ουσία. Ευχαριστώ πολύ για τα τόσο πλούσια σχόλια. Βεβαίως, με χαρά ε, σημειώνουμε τις ε, ε, προτάσεις, ε, γιατί τη στρατηγική μας ε, την αναπτύσσουμε σε τρεις άξονες καταναλωτές, παραγωγή και ποιότητα. τα αναφέρατε λοιπόν συστηματικά στις παρεμβάσεις σας. Καταναλωτές λοιπόν. Θέλουμε οι καταναλωτές να τρέφουν εμπιστοσύνη προς την ιστορική αγορά και να βλέπουν ότι γίνονται σεβαστές και ελευθερίες τους. Αυτό το βλέπουμε λοιπόν και στην έννοια της ε, ισότιμης πρόσβασης που έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας γιατί σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να στερείται κανείς της ε, προσβάσεως λόγω της ε, κατοικίας του ή να έχει τιμή που δεν τον ικανοποιεί. Θέλουμε λοιπόν ισότιμη πρόσβαση. Επίσης, ισότιμη πρόσβαση και στον ανταγωνισμό με βάση τους παρόχους που θα πρέπει να συμμορφώνονται εξίσου. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν η πρόσβαση και το αναφέρατε και εσείς στην, στην παρέμβασή σας για, τις, ε, για την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη διανοτική παραγωγή και ιδιοκτησία και το πόσο μπορούν να έχουν ε, αυτήν την ε, προστασία. Έτσι λοιπόν και η πτυχή του καταναλωτή και η πτυχή της ισότιμης πρόσβασης έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αναφέρατε επίσης σε νεοφύης επιχειρήσεις. Συζητάτε βέβαια και τις νεοφύης αλλά και τις ενισχυόμενες, τις λεγόμενες scale-ups, γιατί με νεοφύης δεν έχουμε τόσο πρόβλημα όσο με scale-ups, δηλαδή αυτές οι οποίες ενισχύουν την ε, ε, παρουσία του σε μια αγορά. Και εκεί έχουμε να κάνουμε ιδιαίτερα με τον προβλημασμό του σχετικό με το ΦΠΑ, με το εταιρικό δίκαιο, με τη χρηματοδότηση, το κόσμο και τη χρηματοδότησή του, το ε, κεφάλαιο διακινδυνεύσεως και ούτω καθεξής. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν αυτό. Και η απόδοση που οπωσδήποτε μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο χάρη σε μια αποτελεσματική ε, νομοθεσία. Αυτό το ανέφερε θα το αναφέρει και η Κέρσταν σε λίγο. Η κοινοποίηση ωστόσο είναι πολύ σημαντική ως παράδειγμα για την ε, ε, διάθεση των αγαθών και την απάλληψη των φραγμών. Βλέπουμε ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες όλο και περισσότερο είναι παρόντα σε ε, ε, έχουμε μια μεικτή οικονομία πλέον, δηλαδή προσφέρονται ταυτόχρονα αγαθά και προϊόντα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Έχουμε να κάνουμε με θέματα που μπορεί να είναι τοπικά, αλλά μπορεί να μην είναι και τοπικά, γιατί αν έχουμε έναν ε, κάτοικο της Μαδρίτης που ταξιδεύει στο, στην Τσεχία, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα της εφαρμογής Φερρυπίν του Uber γιατί δεν ισχύει εκεί και δεν επιτρέπεται πρέπει να αντιμετωπίσουμε το, τη στρέβλωση αυτή στην αγορά μπορούμε να ενθαρρύνουμε την απασχόληση αν και, αν και υπάρχει ταυτόχρονα και ο κίνδυνος του καλυσβαντισμού εις βάρος της ε, ε, απασχόλησης πρέπει να δούμε τα θέματα των, ε, της ευθύνης της ασφάλισης, της αξιολόγησης και όλα αυτά πριν καταλήξουμε σε προτάσεις συγκεκριμένε για όλο τον τομέα. Για δε τον ιό της απορρίθμισης και της επιχρήσωσης. Όσο, πιο, όσο πιο πολύ ε, εναρμόνιση, όσο πιο πολύ μάλλον αμοιβαία αναγνώριση έχουμε, τόσο πιο πολύ εναρμόνιση και καλύτερη λειτουργία της αγοράς. Εκεί που μπορεί να βλέπετε στις υπερβολικές ρυθμίσεις έχουμε να κάνουμε με πιο ε, ολοκληρωμένη αγορά. Και βέβαια αντίστροφα μπορεί οι τεχνικές λεπτομέρειες να μην καλύπτονται. Και βέβαια μπορούμε να έχουμε νομοθεσία λιγότερο τεχνική, λιγότερο λεπτομερή. Αυτά Στηριζόμεθα βέβαια στη δική σας υποστήριξη ως προς τον προσδιορισμό επακριβώς του φάσματος το οποίο θα πρέπει να υπάρχει αυτή η, δια... η διάταξη από την απορρίθμιση μέχρι και την πιο λεπτομερή ρύθμιση σε όλο αυτό το φάσμα που βέβαια δεν πραγματευόμαστε και με τους ε, επαγγελματίες πάντα του κλάδου και η τάση μπορεί να είναι προς την απορρίθμιση περισσότερο αλλά μερικές φορές υπάρχει και εναρμόνιση των ρυθμίσουν και όπως και να έχει θα πρέπει να είμαστε σε επαφή μαζί σας πάντα. Και μια και μου έχει υποδειχθεί να το επισημαίνω κάθε φορά, το ξαναλέω, δεν θα ξανανοίξει η, υπηρεσία, η οδηγία για τις υπηρεσίες. Δεν θα χρειαστεί να ξανανοίξει η οδηγία για τις υπηρεσίες. Πολύ σύντομα. Θέλω και εγώ να σα ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Ήταν πολύ επικοδομητική. Και θα ήθελα επίση να σα ευχαριστήσω για την υποστήριξη που εκφράσατε στι προτάσει μου. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα η Επιτροπή μα μπορεί να πράξει αυτό το οποίο εννοεί και θέλει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να υποταχθούμε στην ιδέα ότι κάποιοι θεωρούν ότι είναι υπερβολικά ήπια η πρόταση επιτροπής και όχι αρκετά σκληρή και να παρετηθούμε σε αυτό. Μπορούμε να την καταστήσουμε πιο σκληρή. Έχουμε να κάνουμε με προτάσεις οι οποίες μπορεί να είναι ε, δημοφιλείς αλλά όχι απαραίτητα και ε, λαϊκιστικές προτάσεις που μπορεί να είναι λειτουργικές και πραγματοποιήσιμες και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι κέρια σημασία η υποστήριξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή με βάση και την έκβαση της ακρόασης και αυτή πρέπει να είναι η εστίαση που θα αξιοποιήσουμε και σε σχέση και με τον παραγωγό γιατί ο παραγωγός κάποια στιγμή είναι καταναλωτής και έτσι άρα είναι, άρα είναι κλειστός αυτός ο κύκλος. Για το διαβατήριο των υπηρεσιών αναζητούμε μια εναρμόνιση προκειμένου να εξασφαλίσουμε κοινού κανόνε διοικητικού, γραφειοκρατικού χαρακτήρα κτλ. Σε αυτό περιορίζομαι εγώ. Οι βασικέ ιδέε θα πρέπει να ισχύουν για του πάντε και από εκεί και πέρα α κερδίσει ο καλύτερο, μια και στον ανταγωνισμό οι ικανότητε και η αξία είναι αυτοί που θα προσδιορίσουν είναι αυτές που θα προσδιορίσουν ε, τον νικητή σε μια σχέση ανταγωνισμού. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την πολύ καλή συνεργασία και εύχομαι κάθε επιτυχία. Um, σας ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Να σας θυμίσω ότι η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών, μάλλον η εξέταση είπαμε 25 Ιανουαρίου και η υποβολή τροπολογιών μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου με δημόσια κρόαση 23 μάλλον 22 και 23 ε, Φεβρουαρίου. Περνάμε τώρα στην εξέταση εκθέσεων, νομοθετική εξέταση, όπου πρέπει να καλύψουμε τρία διαφορετικά θέματα σήμερα. Πρώτη είναι η έκθεση της Επιτροπής για τις κατεξοδότησης πράξεις για τον κανονισμό περί προϊόντων ε, του κατασκευαστικού τομέα. Μετά έχουμε μια ώρα. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο τώρα στην Φούλβια Ραφαέλη από τον DG Grow για να μιλήσει για τον κανονισμό για τα προϊόντα του κατασκευαστικού τομέα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και καλημέρα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσω την έκθεση της Επιτροπής για τις κατεξιδότητες συναρμοδιότητες στο πλαίσιο του κανονισμού ε, για τα προϊόντα του κατασκευαστικού τομέα. Στην έκθεση αυτή θεωρούμε πως αυτές οι αρμοδιότητες ασκήθηκαν εντός της εντολής που μας είχε δοθεί για και αυτό για τρεις ε, κύριους λόγους. Καταρχήν, οι νέα κατεξοδότηση πράξεις που ισχύουν σήμερα αφορούν τομείς που είναι, εντοπίζονται στο άρθρο 60 του κανονισμού και ανταποκρίνονται σε ρυθμιστικές ανάγκες που τις εντόπισαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς και σέβονται τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Δεύτερον, όταν προετοιμάζαμε τις καταξιδότητες εν ε, εργαστήκαμε σε πλήρη διαφάνεια, ήρθαμε σε επαφή με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες και τους ενδιαφερόμενους φορείς, στην Επιτροπή αυτή, το Κοινοβούλιο των ημερών τακτικά για τις δραστηριότητές μας, και σας καλέσαμε και πολλές φορές να συμμετέχετε στις συνεδριάσεις μας. Σε τρίτη παρατήρηση, στη διάρκεια της περίοδου αντιρρήσεων δεν λάβαμε ποτέ καμιά ένσταση ούτε από το Ευρωκοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προσέχουν οι συνομοθέτες αυτές τις κατεξοδότητες συμπράξεις. Αντιθέτως, τακτικά λάβαμε ενημερώσεις και αιτήματα για επιπλέον πληροφορίες για την τεχνική πτυχή όλων αυτών και η Κομισιόν είναι έτοιμη να συνεχίσει αυτό το διάλογο και να ε, ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες. καθώς και να προβεί στα όλα τα απαραίτητα, στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων. Τέλος, η έκθεση επιβεβαιώνει το γεγονός ότι θα χρειαστεί παράταση των κάτω πράξεων και ε, θα συνεχίσουμε να χρειαζόμαστε αυτές τις αρμοδιότητες και για το μέλλον, κυρίως έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την ταχεία τεχνική πρόοδο και τις εξελισσόμενες ανάγκες της βιομηχανίας των ε, ε, κατασκευών. Χρειαζόμαστε καθημερινά νέα είδη ε, κατά εξουσιοδότηση πράξεων σε σχέση με το άρθρο 60. Για να ανταποκριθούμε στην ε, έτοιμα να απευθυνθούμε στα τεχνικά και ε, αναπτυξιακά προγράμματα. Ιδιαίτερα αυτές οι πράξεις πρέπει να Μάλλον θα πρέπει να αρθούν οι πιθανοί φραγμοί και να ελαφρυνθούν ε, το διοικητικό άχθος ε, στον τομέα των κατασκευών. Από αυτές τις βάσεις, τα πρώτα πέντε χρόνια εφαρμογής, η Κομισιόν θεωρεί πως είναι απα, απολύτως απαραίτητο να διατηρηθούν αυτές οι αρμοδιότητες και για το μέλλον. Επίσης θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να επιβεβαιώσω ότι η Κομισιόν εργάζεται για μια έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού σε σχέση με τα προϊόντα του κατασκευαστικού τομέα. Η έκθεση αυτή θα είναι έτοιμη το 2016 και ζητούμε να ληφθεί υπόψη από τον συνομοθέτη ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή αυτού του πολύ σημαντικού νομικού κειμένου για την εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ. Είναι λίγο ατυχές που ο εισηγητής δεν είναι εδώ. Θα μιλήσει κανείς εξ ονόματος της, εισηγητρίας. Όχι. One question that I believe has been asked by a number of members is issues to do with fire safety. Does the Commission want to come back on what your current thinking? Fire Είναι άλλο θέμα αυτό που είπα για την ασφάλεια. Ναι, θα έλεγα ότι είναι αρκετά διαφορετικό θέμα, επί το οποίο βεβαίως εργαζόμαστε και ερευνούμε, αλλά δεν βρίσκεται στο πυρήνα αυτής της συζήτησης. so it is not part of this delegated delegated act, but will come back on future acts, Είναι και αυτό για κατεξοδότηση πράξη, αλλά θα επανέλθουμε στις μελλοντικές, έτσι. Okay. Ναι, ναι, θα μπορούσε όντως να γίνει κάτι τέτοιο. Um, the next issue is on registration of motor vehicles. Τώρα, επόμενο θέμα, η καταχώρηση καταγραφή των οχημάτων με κινητήρα. And I understand Johanna Jaska, Was anybody else in the Commission here to speak about the? So I understand Barbara Bonbisuto is here, is that correct? Barbara, would you like to Μπάρμπαρα. On the η Μπάρμπαρα για αυτό το θέμα. On registration of motor vehicles in the e Μάλιστα, πρόκειται για τη τρέχουσα κατάσταση. Ευχαριστώ που φάλατε το θέμα αυτό. Η Στην ημερήσια διάταξη η Κομισιόν αποδίδει μεγάλη σημασία στο θέμα Στόχος είναι να αφαιρεθούν ε, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες όταν προσπαθούν να καταχωρήσουν ένα έγγραφο που ήδη είναι καταχωρημένο σε άλλο έγγραφο. Και αυτά εμπόδια είναι ανάμεσα στα 20 κύρια εμπόδια της εσωτερικής αγοράς. Η Κομισιόν λοιπόν υιοθέτησε μια πρόταση στις 4 ε, Απριλίου 2012. Έκτοτε συνεχίζονται διαπραγματεύσεις και το κύριο εκρεμές συζήτημα στο επίπεδο της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου είναι το περίφημο άρθρο 3, δηλαδή η ημερομηνία της ε, καταχώρησης. Έχει σημειωθεί πρόοδος, κάποια πρόοδος, διότι στη τελευταία συνεδρίαση της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου κατέστησε σαφές ότι τώρα όλα τα κρατημέλη είναι πεπισμένα πως το άρθρο 3 θα πρέπει να μείνει εντός της προτάσεως, αλλά ότι εξακολουθεί να υπάρχει η συζήτηση ε, όσον αφορά τη σύνταξη του άρθρου 3. Τώρα, μια συμβιβαστική ε, είναι υποσυζήτηση, σύμφωνα με την οποία το κύριο κριτήριο θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι η κατοικία του κατόχου του πιστοποιητικού καταχώρησης. Ε, αυτό θα είναι το βασικό κριτήριο για την υποχρέωση να μεταφερθεί η καταχώρηση. Ωστόσο, κατέστη σαφέ ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια ευελίξια και κάποιο, κάποια κριτήρια για εξαίρεση αναπαραίτητα, τα οποία θα βασιστούν στην έννοια της κύριας χρήσης του οχήματος. Κάτι το οποίο, μάλιστα, εισάγεται και στην έκθεση του Κοινοβουλίου. Ξεκολουθούμε να το συζητάμε. Για να δούμε αν θα ήταν αυτό αποδεκτό από όλα τα κρατημέλη και από την άποψη της, ε, πλευρά της Κομισιόν είμαστε έτοιμοι ώστε να βοηθήσουμε την επίτευξη συμβιβαστικής λύσης. Προφανώς όσο μια τέτοια λύση είναι σύμμορφη προς την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, το Δικαστήριο και την νομολογία, ε, αλλά όπως είπα τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση όπου οι συζητήσεις είναι επικοδομητικές ε, θα πρέπει να γίνει μια επόμενη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας τον Ιανουάριο ώστε να ε, δρομολογηθεί η συζήτηση και να ξαναρχίσουν οι συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, Ντίτε. Θες να πεις κάτι, πεις η συγγήτρια και μετά η Μαρία Γκραπίνη. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι και καινούριο το πρόβλημα. Ήδη το έχουμε επισημάνει εδώ και χρόνια. Μάλιστα ως ένα από, τα, από τους πιο σημαντικούς μη δασμολογικούς φραγμούς για τον πολίτη και τον καταναλωτή. Χαίρομαι που μας ενημερώνει για τις εξελίξεις από το Συμβούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημειώνω ότι έχει δουλέψει σκληρά για το θέμα αυτό από το 2012 ήδη όταν πρότεινε νέο κανονισμό και με χαρά Ακούω νέε προτάσει από την Επιτροπή φυσικά. Θα έπρεπε σήμερα να έχουμε εδώ εκπρόσωπο του Συμβουλίου πάνω απ' όλα. Με χαρά σημειώνω κινητικότητα σε επίπεδο Συμβουλίου. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτερα από ό,τι μέχρι τώρα. Οι διαφορές δεν είναι τόσο βαθιές ώστε να μην μπορούμε να βρούμε ε, σημείο σύγκλησης με τους, ε, μεταξύ των συνομοθετών. Έτσι λοιπόν και ενώ είμαστε έτοιμοι να δώσουμε απαντήσεις σε ένα από τα κύρια μελήματα και ανησυχίε των πολιτών μας φαίνεται το Συμβούλιο, εμείς και η Επιτροπή φαίνεται το Συμβούλιο δεν είναι διατεθειμένο να πράξει το ίδιο. Ελπίζω σε μεταγενέστερε συνεδριάσει επαφέ με την Ολλανδική Προεδρία να μπορέσουμε να δώσουμε ε, ουσιαστικά ελπίδα για του πολίτε και καταναλωτέ. Μαρία Γκραπίνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, λυπάμαι για την καθυστέρησή μου, γιατί είχα και άλλες συζητήσεις να κάνω, λοιπόν, για το θέμα μας. Είδα ότι υπάρχει επιστολή των συναδέλφων από τον Απρίλιο του 2014. Δεν ξέρω αν δόθηκε απάντηση σε αυτή την επιστολή. Η Κομισιόν λέει ότι έγιναν, σημειώθηκαν πρόοδοι, ναι, μάλιστα, αλλά το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάσισε και στο Βέλγιο και μερικές άλλες χώρες φαίνεται ότι δεν εφαρμόζονται ομοιόμορφα οι αποφάσεις αυτές. Αν έρθει να με επισκεφθεί ο άντρα μου από τη Ρουμανία στο Βέλγιο με αυτοκίνητο πρέπει αμέσως να καταγραφεί με κίνδυνο να κατασχεθεί το όχημα. Να, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Θέλουμε να λειτουργήσει πράγματι η εσωτερική αγορά, αλλά να, ένας τεράστιος φραγμός. Δεν ξέρω αν μπορεί να μου απαντήσει η καμισιόν σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Έχει υπάρξει πρόοδος αλλά μου έχουν πει πολλές φορές ότι το θέμα των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων από χώρα σε χώρα είναι κάτι πολύ ακριβό στην Ευρώπη, πολύ παραπάνω από ό,τι στις Ηνωμένε Πολιτείες. Παραδείγματος χάρη μια εταιρεία μπορεί να έχει περισσότερα έξοδα αν διακινεί αυτοκίνητα στο νότο το χειμώνα αντί στο βορρά το καλοκαίρι. Επίσης γνωρίζω ότι τα τρομερά γεγονότα στο Παρίσι αφορούσαν επίσης ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο από το Βέλγιο. Θα ήθελα να είμαστε 100% βέβαιοι ότι η πληροφόρηση που έχουμε για το ποιος βρίσκεται σε ένα αυτοκίνητο, είτε είναι νοικιαζόμενο είτε όχι, είναι επαρκής και ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας θα μπορούν ανα πάσα στιγμή να γνωρίζουν όπως γίνεται με τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σε μία χώρα, τι γίνεται και με τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν μεταξύ χωρών. Πρέπει λοιπόν να είμαστε βέβαιοι ότι η ασφάλεια καλύπτεται. Ξέρω ότι θεωρητικά υπάρχουν συστήματα ελέγχου στην πράξη όμως ίσως να μην είναι. Μήπως η Καμισιόν θέλει να προσθέσει τίποτα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι Όλα αυτά τα ξέρουμε, τους στόχους δηλαδή, τη νομική σαφήνεια, ασφάλεια για τους πολίτες, για να διευκολύνουν τη ζωή των επαγγελματιών, αλλά επίσης να διασφαλίζεται ότι ό,τι και να προτείνουμε θα είναι εύκολα εφαρμόσιμο και δεν θα υπονομεύει με κατά κανένα τρόπο τη δυνατότητα των χωρών μελών να εφαρμόζουν τους κανόνες κυκλοφορίας. Ίσως είναι και αυτός ένας από τους λόγους για τους οποίους μία απόφαση που να είναι αποδεκτή από όλους και αεροστεγής είναι πολύ δύσκολο να κατορθωθεί. Ωραία. Κοιτάξτε, η επίτευξη ενός στόχου και η διασφάλιση ότι έχει πράγματι εφαρμοστεί είναι, δεν είναι κάτι προφανές. Καθαρισμός μάλλον ενό. στόχου. Ας περάσουμε όμως το επόμενο θέμα, ας περάσουμε. Ας περάσουμε. Ευχαριστούμε την κυρία Κέρστεν Ζουρνά. από την Ουδού Γκρόου που θα μας μιλήσει για ορισμένες περιπτώσεις παραβιάσεων. Είναι συνέχεια μια συζήτηση στην ανταλλαγή απόψεων μάλλον που είχαμε με την Καμισιόν για τις περιπτώσεις παραβιάσεων και εκείνη η πρώτη ανταλλαγή απόψεων είχε γίνει τον περασμένο Οκτώβριο. Το κύριο θέμα είναι να δούμε σε ποιους τομείς γίνονται πιο συχνά οι παραβιάσεις ή ποιος είναι ο τύπος των συχνοτέρων παραβιάσεων και να πάρουμε και μαθήματα από τις περιπτώσεις αυτές. Είναι μέρος της ευρύτερης συζήτησης βέβαια για την στρατηγική για την ενιαία αγορά για την οποία μιλούσαμε από το πρωί. Δυστυχώς μερικοί έπρεπε να φύγουν γιατί υπάρχουν ψηφοφορίες και σε άλλες επιτροπές, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μας ακολουθούν εν πνεύματι. Και φυσικά την έκθεση αυτή θα την κυκλοφορήσουμε και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη πλήρη και αναπληρωματικά. Το θέμα είναι βέβαια πώς να βοηθήσουμε να χυθεί άπλετο φως σε αυτό το θέμα των παραβιάσεων. Δίνω λοιπόν το λόγο στην Κέρστεν Ζουρνά. Ευχαριστώ πράγματα. Την προηγούμενη φορά που ήρθα δεν υπήρχε ενιαία στρατηγική. Τώρα υπάρχει αλλά το να εφαρμοστεί είναι το θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να σας δείξω με μία διαφάνεια, μία και μοναδική, τον κύκλο της συμμόρφωσης. Well, While we are trying to get it on the screen, the making it work. Just take some time to get it on the screen, if we can, and to get the lights down. there it is. Can we get the lights down a bit? Για σβήστε τα φώτα παρακαλώ. Λοιπόν, η εφαρμογή σημαίνει ότι υπάρχουν κανόνες. Όχι τα φώτα σβήστε είπα παρακαλώ, γιατί αλλιώς δεν βλέπουμε με φώτα. Σβήστε τα φώτα για να βλέπουμε. Ου, τα φώτα. Ξαναλέω, σβήστε τα φώτα για να βλέπουμε καλύτερα. τα φώτα. Βέβαια έτσι δεν θα μας βλέπουν οι κάμερες της τηλεοράσεως, αλλά πρέπει και εμείς να βλέπουμε. Ναι, ναι. Φώτα. Can I Καλά θα σας τα πω προφορικά λοιπόν. Εδώ βλέπετε έναν κύκλο ζωής κάποιου κανόνα. Αρχίζει με την πρόταση της Καμισιόν, εγκρίνεται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη. Και εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Οι υπουργοί επανέρχονται στις πρωτεύουσες των και ξεχνάνε τι ψήφισαν. Το πρώτο λοιπόν είναι πώς να καταγραφούν όντως οι οδηγίες στα κράτη-μέλη τα οποία έχουν βελτιωθεί στον χρόνο που χρειάζονται για τη μεταφορά. Αλλά υπάρχει και το θέμα της ποιότητος της μεταφοράς. Βρίσκουμε νομοθεσίες που δεν τα καλύπτουν όλα οι νομοθεσίε που τα καλύπτουν όλα πέραν και από την, τα προβλεπόμενα από την οδηγία. Αυτό λέγεται gold plating, επιχρήσωση. Και επομένως είναι τόσο μεγάλη η ποσότητα των εγγράφων που δεχόμαστε για επαλήθευση που δεν είναι δυνατόν να τα διαβάσουμε όλα. Έπειτα. Αυτή τη στιγμή δημιουργούμε ένα εργαλείο αναλύσεως δεδομένων που να μας επιτρέπει σε καμιά εβδομάδα να διαπιστώνουμε αν η νομοθεσία που εγκρίνεται έχει μεταφερθεί, καλύπτει τα πάντα, αλλά και την επιχρήσωση που ίσως έχει γίνει πέρα από αυτά που είχαμε προβλέψει εμείς. Έτσι θα γνωρίζουμε πολύ γρήγορα τι ισχύει, αν είναι υπερβολικό ή όχι αυτό που ισχύει και αυτό χωρίς να χρειάζεται να περιμείνουμε μέχρι να εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα. Όταν έχει μεταφερθεί ένα νομοθέτημα αρχίζει το θέμα της εφαρμογής. Εφαρμογής και από τους πολίτες και από επιχειρήσεις, από ιδιώτες δηλαδή και από τις δημόσιες αρχές. Ε, βλέπουμε λήψεις και στα δύο τμήματα. Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες λένε δεν ήξερα ότι είχα αυτό το δικαίωμα, δεν ήξερα, δεν ήξερα ότι είχα αυτή την ευκαιρία διότι ε, δεν το βρίσκουν στην εθνική νομοθεσία. Δεν υπάρχει επίγνωση. Καινούργιες επιχειρήσεις πολλές φορές δεν γνωρίζουν πού να βρουν την νομοθεσία που μπορεί να ισχύει για τη δραστηριότητά τους. Και επίση υπάρχουν οι κρατικές αρχές που πρέπει να διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι κανόνες επιτήρησης εποπτείας της αγορά δεν το έχουν για προτεραιότητα. Κατανοητό αυτό είναι μέρη. Δεν υπάρχουν δηλαδή τα εργαλεία σήμερα που να διασφαλίζουν ότι αν ανακαλυφθεί ένα ένα νομοθετικό προϊόν θα εφαρμοστεί ομοιόμορφα παντού. Δεν έχουμε τέτοια εργαλεία δοκιμής. Και εδώ έρχεται ο ρόλος της στρατηγικής για την ενιαία αγορά. Να διασφαλίζει δηλαδή ότι οι αρχές είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, έχουν βάλει την πρίζα και έχουν τα μέσα να εφαρμόσουν. Πολλά βέβαια προϊόντα που δεν προβλέπονται από την νομοθεσία προέρχονται εκτός ένωσης. Οι οικονομικοί παράγοντες δεν γνωρίζουν πάντοτε τα πράγματα. Δεν γνωρίζουν. Άρα πρέπει να γίνει ακόμα πιο γνωστό και διαφανές τι ισχύει και ποιοι κανόνες πρέπει να εφαρμοστούν ιδιαίτερα για το Digital Single Gateway όπου θα βρίσκουν την πληροφορία που χρειάζονται. Όχι όμως μόνο να βρίσκουν, αλλά να έχουν και τη βοήθεια που χρειάζονται για να καταλάβουν πώς εφαρμόζονται οι κανόνες. Μιλήσατε για τα σημεία single contact. Και εδώ χρειάζεται καλύτερη διασύνδεση. και μετά υπάρχει το τμήμα Smart Enforcement που αφορά τις παραβιάσεις. Και εδώ έχουμε άλλη διαπάνεια. Όταν έχουμε 28 χώρες και 560 εκατομμύρια καταναλώτριους πρέπει να βρούμε έναν έξυπνο τρόπο για να διασφαλίσουμε πώς θα στοχεύουμε τους σπουδαιότερους. Να, εδώ, εδώ βλέπετε την ισχύουσα τάση από το 8 και μετά οπότε και άρχισε η πειραματική φάση διοικητική συνεργασία μεταξύ των μελών υπάρχει 45% μείωση των περιπτώσεων που έχουν διαπιστωθεί. Από χίλιες περιπτώσεις έχουμε φτάσει στις 730. Άρα δουλεύει το πράγμα να ταυτίζεται το πρόβλημα εγκαίρως για να μπορεί να λυθεί εγκαίρως. Όταν μιλούμε για έξυπνη εφαρμογή εννοούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παραβιάσεις για να βελτιώσουμε τη στρατηγική, να αυξηθεί η αποτελεσματικό της δηλαδή. Για τις επενδύσεις θα τα πούμε αργότερα. Αργότερα. Καμιά φορά πρέπει να υπάρχει και κατάργηση ορισμένων κανόνων γιατί θα ισχύσει η αμοιβαία αναγνώριση και τέλος η πολιτική μας δημοσίων προμηθειών μπορούμε να ανοίξουμε τις αγορές των χωρών μελών για τις δημόσιες αγορές. Ένα πρόσφατο παράδειγμα. Η Επίτροπο Αμπιανκόφσκα άρχισε διαδικασίες δίωξης έξι χωρών μελών γιατί δεν είχε εφαρμοστεί σωστά η οδηγία που επέτρεπε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ένα νομοθέτημα μόνο αν είναι αυτός ο μόνος τρόπος επίτευξης του στόχου. Αναλογικότητα δηλαδή. Το περασμένο Ιούνιο εγκρίθηκε αυτό. Τώρα θα σας δείξω μια άλλη διαπάνεια. Οι reasoned opinions που είναι η φάση όπου η διοικητική συνεργασία προσπαθεί να βρει μια λύση όποτε δεν το έχει πετύχει κάποιο κράτος μέλος. Παίρνουμε αυτές τις περιπτώσεις και λέμε στα κράτη-μέλη αν δεν το λύσετε θα σας πάμε στα δικαστήρια. 214 τέτοιες περιπτώσεις έχουμε, reasoned opinions, εμπεριστατωμένες γνωματεύσεις αιτιολογημένες ονοματεύσεις Τις έχουμε αναχώρα και ανατομέα. Αν επιστρέψω ανατομέα, ανατομέα. Εδώ βλέπετε ότι προσπαθούμε να γίνουν όλα αυτά πιο στοχευμένα για το περιβάλλον ας πούμε. 16 περιπτώσεις για την κακή εφαρμογή της οδηγίας της ποιότητας του αέρος. Για επιστρέψτε παρακαλώ στην προηγούμενη διαφάνεια. Αυτή είναι αναχώρα. Εγώ λέω ανατομέα, να, να, ναι, εδώ ανατομέα. Ανατομέα εκείνο το μεγάλο τμήμα πάνω πάνω κλπ. Το γαλάζιο είναι περιπτώσεις που έχουν πάει ήδη στο δικαστήριο και το μπλε ή αιτιολογημένες γνωματεύσεις ή γνωμοδοτήσεις. Έχουμε για τη διαχείριση των αποβλήτων ας πούμε, για τις μεταφορές 10 περιπτώσεις για την νομοθεσία για τις άδειε οδήγηση που αμφισβητούνται. Επίσης για τα μητρώα των αυτοκινήτων έχουμε 20 περιπτώσεις παραβίασης σε διάφορες φάσεις της διαδικασίας. Προσπαθούμε να το λύσουμε. στο θέμα των προσφυγών. 7 οδηγίες για την παραβίαση της ελεύθερης διακίνησης. Τώρα αναχώρα πάλι. Αυτονόητο. Δείχνει ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ χωρών μελών. Και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ άλλων τύπων χωρών μελών. Αυτό για τις παραβιάσεις. Θα επανέλθω μετά όμως για να δω πώς μπορούμε να τα ομαδοποιήσουμε όλα αυτά. Πριν όμως θα ήθελα να προσέξετε κάτι άλλο σημαντικό εργαλείο που έχουμε για την αποφυγή, για καλύτερη μάλλον εφαρμογή η διαδικασία notification γνωστοποίησης. Πρέπει να γνωστοποιούνται όλα τα σχέδια τεχνικής νομοθεσίας πριν εγκριθούν από τα εθνικά κοινοβούλια. Και μπορούν να σχολιάσουν και οι χώρες μέλη και η Καμισιόν και να ζητήσει από τη χώρα μέλος να αλλάξει το σχέδιό της. Είναι ο προθάλαμος αυτός της ενιαίας αγοράς στον προθάλαμο αυτό μπορούμε να αποφύγουμε τη δημιουργία φραγμών πριν αρχίσουν να υπάρχουν. Είναι πρόληψη, πρόληψη, όχι θεραπεία. Πρόληψη. Και αυτή η οδηγία οφείλεται στο κοινοβούλιο σας, διότι το 15 συστάθηκε. And just to give you an idea of how important it is, we have something like 700 notifications. Έχουμε 700 τέτοιε γνωστοποιήσεις από τα κράτη-μέλη το χρόνο. Σχέδια γνωστοποιήσεων, όχι γνωστοποιήσεις. Ε, κατά μέσο όρο η Κομισιόν στέλνει περίπου 17 λεπτομερείς γνωμοδοτήσεις όπου λέει αν εφαρμόσετε το α θα παραβιάσετε το κοινοτικό δίκαιο και 160 σχόλια το χρόνο όπου λένε βελτιώστε την πρόταση. Αλλά όχι μόνο η Κομισιόν και άλλες χώρες μέλη. Είναι ισότιμη διαδικασία λοιπόν. 70 κίτρινες κάρτες από άλλες χώρες μέλη. Και μπορούν οι παράγοντες να συμβουλευτούν αυτό τον ιστότοπο που λέγεται τρεις. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στη συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία γιατί όλοι ξέρουν ότι ό,τι καταργηθεί σε αυτή τη φάση δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στη συνέχεια στην ενιαία αγορά. Επίσης προσθέτω ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μας βοηθάει διότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε εάν μια χώρα μέλος δεν γνωστοποιήσει, ενώ θα έπρεπε να είχε γνωστοποιήσει, τότε αυτό το νομοθέτημα δεν μπορεί να τύχει προσφυγής στο δικαστήριο. Και οι δικηγόροι σιγά σιγά το εκμεταλλεύονται αυτό το παραθυράκι. Τώρα πώς να συνεργαστούμε για να βελτιωθεί η συμμόρφωση με την ενιαία αγορά. Καταρχήν η έγκαιρη μεταφορά, διότι αν εγκρίνει κανείς ένα νόμο στο, στις και δεν φτάσει στα κράτη-μέλη δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε να εξηγήσουμε μαζί την αναγκαιότητα για έγκαιρη μεταφορά. Στη δέσμη που σας στείλαμε υπάρχει κατάλογος όλων των οδηγιών, 114 νομίζω σύνολο, που θα χρειαστούν μεταφορά κατά τη διάρκεια της εντολής σας της θητείας σας. Μπορείτε να μας βοηθήσετε με τις χώρες σας. Ε, μετά υπάρχει το θέμα της κουλτούρας της συμμόρφωσης. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της στρατηγικής της ενίας αγοράς. Στη δέσμη που σας δώσαμε υπάρχει κατάλογος των ανακοινώσεων τύπου που κάνει κάθε μήνα η Κομισιόν όταν που αφορούν ε, παραβιάσεις για τις αιτιολογημένες που σας έλεγα πριν η Κομισιόν δίνει πολλές πληροφορίες και εδώ θα μπορούσατε ίσως να μας βοηθήσετε να μας το πείτε αν μπορείτε είναι δημόσιες αυτές οι πληροφορίες και αν θέλετε μπορούμε να σας στείλουμε και τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο Κάθε μήνα αποφασίζουμε ποιες θα είναι οι παραβιάσεις από τον Ιανουάριο βέβαια και μετά μέχρι και το Δεκέμβριο 12 μήνες και μετά υπάρχει το θέμα της γνωστοποίησης νομοσχεδίων όπου υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ χωρών μελών. Μερικές γνωστοποιούν πολύ και άλλες καθόλου. Μόνο σχολιάζουν. Προσπαθούμε να δούμε τι γνωστοποιήσεις δεν έγιναν, αλλά η διαδικασία αυτή έχει τη φήμη ότι είναι σαλαμοποιητής ή σαλαμοποιήτρια και ότι οι εταιρείε του κράτου μέλους που δεν γνωστοποιούν μπορεί να εμποδίζονται να εξάγουν λόγω της νομοθεσίας που το κράτος μέλος μπορεί να έχει αφαιρέσει κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής φάσης. Επίσης αν θέλουν μπορούμε να κάνουμε να οργανώσουμε εργαστήρια στα κράτη-μέλη, σεμινάρια και εδώ τελειώνει η παρουσίαση του πώς βλέπει η Κομισιόν τη συμμόρφωση την εφαρμογή στην στρατηγική της ενίας αγοράς. Σας ευχαριστώ. Lucy Anderson, and ναι, then Maria Lucy Anderson και μετά η Μαρία. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Μια-δυο ερωτήσεις για γιατί πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση. Θα ήθελα συγκεκριμένα να μου πείτε πώς κατηγοριοποιούνται αυτές οι υποθέσεις εναντί της ε, Γενικής Επιτήρησης της Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Δικαίου γιατί βλέπω να καλύπτεται μόνο το ίμιση του συνόλου των υποθέσεων. Πώς κρίνεται λοιπόν ότι είναι εσωτερική αγοράς ή, ή μη μία περίπτωση. Και ιδιαίτερα στους τομείς όπου έχουμε υψηλά επίπεδα παραβιάσεως. Στο χώρο του περιβάλλοντος το πρόβλημα το έχουμε παγίως και το έχουμε υπογραμμίσει και εμείς και η Επιτροπή μας. Για τον πολίτη δηλαδή και για τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι βασική αξία το περιβάλλον. Δεν μπορούμε να το λησμονούμε και έχει σαφέστατη αρμοδιότητα για κάθε έναν από τους λόγους που μας είναι γνωστοί και σημαντική. Άρα λοιπόν θα ήταν καλό να το κοιτάξει η Επιτροπή μα, έστω και αν δεν είναι απόλυτη αρμοδιότητά ή αποκλειστική αρμοδιότητά τη, γιατί έχουμε με βάση το άρθρο 298 τη συνθήκη ω κοινοβούλιο την αρμοδιότητα να κοιτάξουμε και να στηρίξουμε όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στις ε, παραβιάσεις τη νομοθεσία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό θέλω να μου κάνετε μία ανάπτυξη σχέση με τη διάσταση εσωτερική αγορά, είτε εσεί είτε η συνάδελφοί σας από την νομική υπηρεσία, κυρία Γκραπίνη. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση όντως. Πολύ σωστά λέτε ότι θα πρέπει να ενημερωθεί η κάθε χώρα για αυτές τις πρωτοβουλίες και πολύ σωστά επίσης λέτε ότι αφενός ε, η αρχές πιέζουν ε, οι εθνικές αρχές μέχρι τέρματος της προθεσμίες υλοποίησης των οδηγιών, φτάνουν μέχρι τελευταία στιγμή. Και επίσης η επιτήρηση της εσωτερικής αγοράς δεν φαίνεται να φέρνει πραγματικά αποτελέσματα. Είναι πολλές οι στρεβλώσεις, είναι πολλά τα εμπόδια για τις ε, δημόσιες προμήθειες. Έχει κάνει η Ρουμανία πολλές ε, προσπάθειες γιατί δεν θέλουμε όταν υπάρχουν αμφισβητήσεις ε, στο τέλος μιας διαδικασίας πλειοδοσίας να αμφισβητείται ένας, το αποτέλεσμα ενός διαγωνισμού γιατί κάθε βέβαια προσφυγή απλώς καθυστερεί ακόμη περισσότερο την υλοποίηση. Εγώ που μάλιστα ήμουν και υπουργό την εποχή που είχε προκύψει το ζήτημα αυτό, είχα ζητήσει να επιβάλλονται κυρώσεις στους προσφεύγοντες εφόσον δεν ήταν βάσιμη η ε, αμφισβήτηση και η προσφυγή τους. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι, διότι είναι καταστροφική κατάσταση για τις μικρομεσαίες. Και βεβαίως πρέπει να αποτρέψουμε αυτούς που προσπαθούν να στρεβλώσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Εσείς επίσης στην παρουσία σας δείξατε ότι όσο πιο ανεπτυγμένο σε ΑΕΠ ή και άλλους οικονομικούς δείκτες ένα κράτος, τόσο και πιο υψηλό επίπεδο τήρησης των κανόνων της εσωτερικής αγοράς ε, επιδεικνύει. Πώς θα το εξηγήσετε αυτό? Ευχαριστώ και και για την λεπτομερή ενημέρωση. Δεν είχαμε την ευκαιρία να το κοιτάξουμε λεπτομέρως γιατί έφτασε μόλις εχθές, θα πρέπει να το ξαναδούμε φαντάζομαι. Ιδιαίτερος πάντως βλέπω να έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η έκθεση αυτή που μόλις παρέλαβα έχει και κάποιες ε, κύριες και κέρυες περιπτώσεις. Κυρίες γιατί θα μας επιτρέψουν να αντιληφθούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ε, παραβάσεις και να καταλάβουμε καλύτερα τα προβλήματα. Δηλαδή μπορεί να έχετε κάποιες συγκεκριμένε ε, υποθέσεις ε, που καταλαβαίνω ότι θα σας προβληματίζουν και ίσως είναι δύσκολο να γίνει η επιλογή της υπόθεσης που θα προωθήσετε περισσότερο με την προσφυγή. Πάντως είναι ενδιαφέρον για μας να έχουμε καλύτερη ενημέρωση για τις επιλογές μας, τις πολιτικές, εάν μπορούμε να καταλάβουμε και περισσότερο το λόγο για τον οποίο γίνονται αυτές οι παραβιάσεις. Ένα θέμα σχετικό με την Ελλάδα που έχει τις καλύτερες επιδόσεις και έχει να κάνει με την παράβαση των κανόνων περί αποδόσης της ενέργειας στην οδηγία για τα κτίρια, κατοχώρες επίσης για την αποτελεσματικότητα στη χρήση και την ε, κατεργασία των λιμάτων. Υπάρχει τρόπος να αντιληφθούμε ποιες από τις υποθέσεις αυτές μπορεί να έχουν μεγαλύτερη απήχηση και που μπορούμε περισσότερο ή που θα οφείλουμε περισσότερο να ανησυχούμε. Ή πρέπει να ανησυχούμε για όλες. Υπάρχει κάτι που μπορεί να μας επιτρέψει να αντιληφθούμε εάν ε, φταίει η νομοθεσία ίδια. γιατί βλέπουμε πάντα να υπάρχει συζήτηση για το πότε θα οριστεί η προθεσμία για την υλοποίηση. Το ΔΕΚΙΝΟΒΟΥΛΙΟ πιέζει για, το ταχύτερο, για, το όσο δυνατόν ταχύτερη υλοποίηση. Το ΔΕ Συμβούλιο ε, λέει «Α, όχι, θέλουμε πιο πολύ χρόνο». Έτσι λοιπόν... Πρέπει να δούμε ποια είναι η ισορροπία ανάμεσα και στην ταχύτητα αλλά και στην ποιότητα, βασικά στο να βεβαιωνόμαστε ότι η νομοθεσία που συμφωνούμε και εγκρίνουμε σήμερα δεν θα χρειαστεί τρία-τέσσερα χρόνια για να υλοποιηθεί. Ήδη είχαμε τη Δευτέρα αναφερθεί στο ζήτημα των εκτελεστικών εξουσιών που θα αξιοποιούσε η Επιτροπή από το 2008 σημειώνω για την από ε, για τον αφοπλισμό των όπλων, για την απενεργοποίηση καλύτερα των όπλων. Ε, βλέπουμε όμως ότι αυτό δεν έχει γίνει ακόμη με τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Θα ήταν καλό να γίνει μια συζήτηση και ίσως κάποιος ε, από κάθε ομάδα θα ήταν σκόπιμο να οριστεί ως υπεύθυνος για να, μας, ε, για να παρακολουθεί την υπόθεση. και κυρίως ε, τις συνθήκες πρότασης της νομοθεσίας και υλοποίησης της στη συνέχεια. Ένα σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να κοιτάξουμε με προσοχή είναι το peer-to-peer review, δηλαδή η αξιολόγηση από τους ε, εταίρους. Θέλετε να λάβετε και πάλι το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Αυτό που σας ε, ε, έδειξα πριν με τη διαφάνεια είχε να κάνει με την ουσία της υλοποίησης και τελικά ότι μόνο η πρακτική εφαρμογή επιβεβαιώνει, επικυρώνει ή απορρίπτει μία πρόταση. Έτσι λοιπόν, μέσα από τις ε, διαδικασίες παραβάσεως διδασκόμαστε και για το τι χρειάζεται βελτίωση. Και αυτό ακριβώς εννοούμε όταν μιλούμε για συμμόρφωση και ευφυή επιβολή δηλαδή να μετατραπεί αυτό να, να αναγνωριστεί η διαδικασία και να μετατραπεί σε νομοπαραγωγική βάση και, αρχή. Σε αυτό θα θέλαμε περισσότερη συνεργασία βεβαίως μαζί σας. Η επιβολή, επίσης να λέμε συμμόρφωση και επιβολή. Ε, πρώτα πρέπει να έρθει η συμμόρφωση, το ownership το λεγόμενο, το να αποδεχθεί δηλαδή κανείς τις προτάσεις και στη συνέχεια, εάν δεν λειτουργήσει αυτό, η επιβολή για τις υποθέσεις. Μπορώ να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες, ε, θέματα που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν πιο συγκεκριμένα. Πάντως εμείς κάνουμε μια διαρκή παρακολούθηση και χαρτογράφηση του, της νομολογίας μας, ε, της περιπτωσιολογίας μας, ώστε να εντοπίσουμε πού μπορεί να προκύπτουν ζητήματα και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πάντοτε ε, υπέτειο θεωρείται ένα νομοθέτημα. Μπορεί να υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός ο οποίος γεννά προβλήματα στην επιτήρηση των αγορών, παραδείγματι. Χρειάζεται μια καλύτερη διασύνδεση γιατί έχουμε τις, ε, την νομοθεσία που μερικές φορές χρειάζεται νομοθετικό ε, μέσον. Άρα λοιπόν όταν έχουμε πολλές αρχές διαφορετικές εποπτείας αγοράς, για να λειτουργήσει η σχετική νομοθεσία πρέπει να διευκολυνθεί η ε, επιτήρηση, να εφαρμόζονται πιο σωστά, πιο εύκολα πρώτα απ' όλα οι νόμοι για να εφαρμόζονται πιο σωστά. Εξού και ο κύκλος της ε, συμμόρφωσης για μένα έχει μεγάλη σημασία και δεν πρέπει να τον λησμονούμε. Και εδώ νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό και περιθώριο συνεργασίας για τις δημόσιες προμήθειες και την αποκατάσταση. Νομίζω ότι ένα από τα μέσα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε είναι να βοηθούμε τα κράτη-μέλη εξαντε προκαταβολικά προ-καταβολικά και όχι εξ να συνεργάζονται σε μεγάλες επενδύσεις να εξασφαλίζουν ότι η διαδικασία των προμηθειών τους είναι σωστή, να μην προκύπτουν ως εκ τούτου καθυστερήσεις για τις επενδύσεις, όπως θα προχωρούν οι διαδικασίες για τις προκηρύξεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό νομίζω. Μάλιστα. Υπάρχει απάντηση για την κατηγοριοποίηση που σας ρώτησα νωρίτερα. Κοιτάξτε. Τη συζήτηση αυτή την κάναμε όταν αναπτύξαμε το βαθμολόγιο για, τις, ε, για την αγορά. Ε, η νομοθεσία της εσωτερικής αγοράς είναι οτιδήποτε στηρίζεται σε, νόμιμη βάση, σε νομι, νομική βάση της εσωτερικής αγοράς. Αυτός είναι ο απλός ορισμός. Και νομική βάση της εσωτερικής αγοράς είναι το συγκεκριμένο άρθρο και τα περί αυτό. Άρα έπρεπε κάπου να χαράξουμε μια διαχωριστική γραμμή. Κάπως έτσι το καταφέραμε. Αυτό. Πρόεδρος. Το, φύλλο το φίλο που μας στείλατε, fact shit, είναι κανονικός ο αριθμός των παραβιάζων ένα μήνα. Ο, διαφέρει από μήνα σε μήνα πολύ. είχα πει να σας στείλω για ολόκληρο χρόνο γιατί κάθε μήνα έχουμε αυτό το δελτίο. Κάθε μήνα. Διαφέρει, διαφέρει ο αριθμός, διαφέρει. Έχουμε ακόμη 10 λεπτά πριν το επόμενο θέμα. 18 βλέπω περιπτώσεις εδώ. 18. Για ενέργεια, Ελλάδα, και οδηγία για την ενέργεια, Γαλλία και Ολλανδία για την ενεργειακή αποδοτικότητα, Γαλλία για τα ραδιενεργά απόβλητα, Ελλάδα για την ε, έριψη αποβλήτων στο πόσιμο είδο, Ρουμανία, και λοιπά Όσα γράφει εδώ στο δελτίο. on over reliance on credit ratings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 and Netherlands on the double taxation treaty between the Dutch in the Dutch Japanese tax treaty. Αυτά. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν αυτά πρέπει να το διαβάζει κάθε επιτροπή κάθε μήνα ανάλογα με την εντολή της. Για να γνωρίζει το Κοινοβούλιο τι ακριβώς συμβαίνει. Και αλλιώς να τα διαβάζουμε κάθε φορά πριν από την ψηφοφορία. Μια ιδέα λέω, μια ιδέα, μια ιδέα. Η Καμισιόν. Καταρχήν, ο κατάλογος που έχετε είναι η ανακοίνωση τύπου της Κομισιόν. Αλλά, εάν έχετε δύο λεπτά ακόμα, θα σας διαβάσω εγώ μερικά από τα θέματα που μας γνωστοποιούν τα κράτη-μέλη για νομοσχέδια για να αποφευχθούν εμπόδια. Τα περασμένα πέντε χρόνια εξετάσαμε τις περιπτώσεις των τομέων όπου τα κράτη-μέλη ασχολήθηκαν με την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων, δρόμους, ε, πυρασφάλεια κλπ radio equipment telecommunication packaging and packaging waste biodegradable waste so that you see the, the, the reality of the single Βλέπετε λοιπόν ότι η πραγματικότητα της ενιαίας αγοράς μπαίνει στον προθάλαμο και είναι πολύ διαφανής, πολύ διαφανής. Μεταφράζεται σε όλες τις κοινωτικές γλώσσες και υπάρχει μια πραγματική δυνατότητα ανταλλαγής με τους χώρες μέλη σε αυτό το τρίμηνο μπλοκ. ώστε να καταλαβαίνουν ότι οι Α και Β εταιρείε δύσκολα θα μπουν στην αγορά του μια χώρας γιατί ισχύουν ας πούμε 15 νομοθετήματα για τα ενεργειακά πατά είναι πολύ σημαντικό εργαλείο λοιπόν. Δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά αν μπορούσατε να μας το γνωστοποιήσετε, γιατί αυτό τα εθνικά κοινοβούλια δεν το γουστάρουν. Δεν τους αρέσει. Αν μπορούσατε να εξηγήσετε πόσο θα μπορούσε να βοηθήσει τους πολίτες και τις εταιρείες των χωρών μελών να συμμορφωθούν, τότε θα καταργούνταν πολύ φραγμοί για όλους και όλες. Ναι, έχουμε δύο εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας με αυτό το θέμα. Η μία είναι στρατηγική για την ενιαία αγορά και το άλλο είναι για την απομάκρυνση κατάργηση μη δασμολογικών φραγμών. Ιδίως αυτό το δεύτερο. Και βέβαια και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα μπορούσαμε να εθαρρύνουμε τους δύο αυτούς συζητητές να εξετάσουν αυτά που μόλις είπατε και να δούμε Μήπως μπορούμε να χύσουμε λίγο περισσότερο φως. Επίσης καθώς είπατε, καμιά φορά οι ίδιοι οι κανόνες που ισχύουν στα κράτη-μέλη εμποδίζουν τις εταιρείε να εξαγάγουν. Να εξάγουν. Υπάρχει και αυτό. Δεν σε αφήνω να πουλήσεις. Έτσι δηλαδή μπλοκάρει μια χώρα τις ίδιες της τις εταιρείες. Σημαντικό ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον, αναποδογυρίζει το επιχείρημα. Θα ευχαριστούμε πολύ. Κέρστεν Ζουρνά. Ευχαριστώ είπα. Τώρα. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη αφορά ενημέρωση για τον τριμερή διάλογο σχέση με την ασφάλεια. Ο Αντρέ Φόπ δεν μπορεί να είναι εδώ εισηγητή για... λόγω άλλων δεσμεύσεων. Με χαρά σα ενημερώνω λοιπόν εκ μέρου του πω ύστερα από δυόμιση έτη διαπραγματεύσεω καταλήξαμε σε μια συμφωνία για την οδηγία επιτέλους τη Δευτέρα το βράδυ και θέλω να απευθύνω θερμότατες ευχαριστίες και στον Ανδρέα και στην, στον Ανδρέας και στην ομάδα του, ιδιαίτερα δε την Άστρετη και την Μπίργκετ από τη γραμματεία της ΣΥΜΚΟ που εργάστηκαν πάρα πολύ σκληρά και επίσης και προς τους Σκιώδης, Νικόλα και τα λοιπά, που ξέρω ότι έμειναν μέχρι τις μικρές πρωινές ώρες να συζητήσουν. Συνοπτικά, για τα πρακτικά μας. Αναφέρεται σε διάφορους τομείς η νομοθεσία, καταρχάς την λειτουργία κεντρικών υπηρεσιών, υποδομές, μεταφορά ενέργειας, υγεία, κυβερνοασφάλεια, τράπεζες, κίνδυνοι για, το για την ασφάλεια, κίνδυνοι για τον κυβερνοχώρο και διαδικασίες εγκάρσιες διασφάλισης καθώς και μηχανισμούς ε, συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών πριν να ε, φτάσουμε στην, στην στον του κινδύνου. Σε ψηφιακό επίπεδο τώρα και η Επιτροπή μας και η Ήτρε λένε ότι δεν θέλουν να καλυφθούν από την παρούσα οδηγία οι υπάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών γιατί είναι διαφορετικά τα συστήματα στις 28 χώρες μέλη και αυτό μας ανησυχούσε. Βρήκαμε μια μέγιστη, μια προς τα άνω εναρμόνιση ως λύση και εξαίρεση για τις μικροεπιχειρήσεις. Exposed εκ των υστέρων ε, έλεγχος απαιτείται για να μπορέσουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις να επαληθεύσουν τις προϋποθέσεις, να ορίσουν τις προϋποθέσεις ασφαλείας, αλλά μετά να γίνεται και εκ των υστέρων η αξιολόγηση της ασφάλειας, ώστε να ξέρουμε ότι υπάρχει η ανάληψη της ευθύνη από την επιχείρηση στο κατάλληλο επίπεδο χωρίς να επιβαρύνεται υπερβολικά με προϋποθέσεις και όρους λειτουργίας. Υπάρχουν κάποια στοιχεία δηλαδή τα οποία δεν καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής, ε, αλλά τα ηλεκτρονικά, ε, το ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές πλατφόρμες κτλ. θα ανήκουν ε, στο πεδίο εφαρμογής. Πάροχοι υποδομών υπάγονται επίσης και άρα είναι σαφείς οι γραμμές και για την υποχρέωση ε, λογοδοσίας. Ε, Σεφέστερη ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ε, κρατών μελών, συντονιστές, μέσω της ενίσα γίνεται ο συντονισμός. Επίσης, υιοθετείται ελπίζουμε από το Συμβούλιο, μια και το κείμενο βρίσκεται τώρα υπό επεξεργασία από τους νομι, νομομαθείς και τις νομικές υπηρεσίες, ένας μήνας για την ε, μεταφορά και έξι μήνες για την ανάπτυξη της κρίσης, των κρίσιμων υποδομών. Ευχαριστώ όλους ε, τους εμπλακέντες και το λόγο θα λάβει ο Νίκολα για να κάνει την αξιολόγηση. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ανδρέα Σφά που δεν είναι εδώ, αλλά φαντάζομαι ότι θα του μεταφερθεί η ευγνωμοσύνη μου και, και εσένα βεβαίως που τον εκπροσώπησες για να παρουσιάσεις τα αποτέλεσματα του τριμερούς, του τριμερούς διαλόγου με την ε, Λουξεμβουριανή Προεδρία και την Επιτροπή χάρη στην οποία μπορέσαμε να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα για τα δίκτυα σε μια χρονική στιγμή όπως η παρούσα ήταν πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία μπορεί να μην επιτύχαμε όλους τους στόχους αλλά πρέπει ιδιαίτερα να τονίσουμε ότι εξασφαλίσαμε τον ένα στόχο δηλαδή την καλή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών τη συνεργατική σχέση και στη συνέχεια μια διαδικασία η οποία θα επιτρέψει στον Ευρωπαίο πολίτη και τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης όπως και τα ΕΟΥΣ, εθνικούς θεσμικούς φορείς, μια πολύ καλή συνεργασία για την ενίσχυση της ασφάλειας των δικτύων. Ευχαριστώ πολύ και την Πρόεδρο και τον εισηγητή βέβαια και τους και όδης που συνεργάστηκαν. Εγώ ανέλαβα ως βουλευτής τον Ιούλιο του 2014 και ήταν η πρώτη, ε, το πρώτο θέμα με το οποίο ασχολήθηκα ως ε, νέος βουλευτής και μάλιστα υπό Ιταλική Προεδρία. Χρειάστηκε ένας χρόνος και ξέρω ότι έχει ξεκινήσει από πιο παλιά ακόμη το θέμα, άρα αποδεικνύεται ότι ήταν πολύ περίπλοκο ζήτημα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να καταγράψουμε και φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό σημείο με τη συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ. Completely agree. Συμφωνώ, συμφωνώ απολύτως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο με πολλές προεδρίες και πολλή δουλειά που έγινε από διάφορες προεδρίες. Ελπίζω λοιπόν ε, τώρα οι κρίσιμες υποδομές να είναι πιο ασφαλείς ε, στην Ευρώπη. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η μείωση των εμποδίων που υπάρχουν. Ξέρω πως η εισηγητής είναι σε μια άλλη επιτροπή και ψηφίζει. Πώς μπορεί κάποιος να τον φέρει για να προχωρήσουμε λίγο. Και έχει τρία λεπτά. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Um, I know there's some big votes happening in other committees, which is why a number... Δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες επιτροπές. Φεύγουν εδώ πέρα οι βουλευτές για να πάνε αλλού. 321, we're going to start. 3824, θα ξαναρχίσουμε. Ή τα 3-2. Λοιπόν, εδώ είναι παρουσίαση μιας μελέτης. Μιας μελέτης λέγω για τη μείωση των φραγμών και του κόστους για τις εταιρείες στην ενιαία αγορά. για να έχουμε στοιχεία για την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για τις μη, τους μη δασμολογικούς Οι συντάκτες της έκθεσης Σαν Jones, Μαρκ Godolf από το London School of Economics έχουν έρθει για να μας παρουσιάσουν τη μελέτη των. Αρχίστε μαζί γιατί οι συγητές πρέπει να πάνε αλλού για να ψηφίσουν. Αλλά ακούτε και από τους παπαγάλους ακούνε, δεν στεναχωριέστε. Υπάρχει και η αναμετάδοση. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Yes. Πρόκειται για μια σύνοψη, μια, μια σύνοψη μιας εκτεταμένης μελέτης για το κόστος και τους φραγμούς ε, στην ενιαία αγορά και τι σχέση έχει αυτό με το πρόγραμμα το, της πολιτικής ε, που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Θα σας ε, πω λίγο πώς μπορείτε να σκέφτεστε Να σας πω λίγο το ιστορικό με τα πώς μετράμε τους φραγμούς και το κόστος πώς ευθυγραμμίζονται αυτά με τις προτεραιότητές μας και τέλος τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε περαιτέρω τους φραγμούς και το κόστος παρακαλώ Ο στόχος εδώ της πολιτικής είναι να μειωθούν οι φραγμοί στην μακροολοκλήρωση και να μειωθεί το κόστος για τις επιχειρήσεις. Έτσι αυξάνεται η συνολική ευημερία καθώς αυξάνεται η παραγωγικότητα σε ολόκληρη την οικονομία Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο ωφελεί μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά την αγορά ολόκληρη. Δεν θέλουμε λοιπόν να διευκολύνουμε μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά οι επιχειρήσεις θα διευκολυνθούν να ανταγωνιστούν σκληρότερα και εντονότερα. Κοιτάξτε, φραγμή και κόστος. Το ίδιο πράγμα είναι υπό μια έννοια, δηλαδή οι φραγμοί μεταφράζονται σε κόστος. Και αν υπήρχε ένας φραγμός ο οποίος φαίνεται αδιάβατος για μια επιχείρηση, το κόστος είναι ουσιαστικά ότι δεν ξεκινάει κανείς μια επιχείρηση σε αυτό το κράτος μέλος. Οπότε είναι όπως σας είπα συχνά ταυτόσιμα αυτά ο φραγμός και το κόστος αλλά θα πρέπει να δούμε φραγμούς που δημιουργούνται από χαρακτηριστικά της αγοράς ή ρυθμιστικούς φραγμούς που δημιουργούνται από την νομοθεσία. Οι φραγμοί της αγοράς περιλαμβάνουν και τις αποτυχίες της λεγόμενης της αγοράς και τις προτιμήσεις των καταναλωτών, διαφορές σε γλώσσα και έθιμα ισχύς της αγοράς, κάτι το οποίο είναι προβληματικό σε κάποιες αγορές και το θέμα της ρύθμισης ε, που προσπαθεί να δει τους φραγμούς. Και βέβαια η ρύθμιση έχει όπως είπαμε έναν δίτο ρόλο. Μια φορά πράγματι εκφράζει τις διαφορές μεταξύ χωρών αλλά μπορεί να εμποδίσουν και την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς και να αυξήσουν τους φραγμούς ε, και το κόστος. Αυτό θα το λέγαμε μια ρυθμιστική αποτυχία και ένας λόγος ε, γι' αυτό είναι πως οι προτεραιότητες δεν είναι σαφείς, δεν έχουν σκεφτεί σωστά τον αντίκτυπο και οι συνέργειες με άλλους τομείς πολιτικής δεν έχουν εξεταστεί και εδώ πέρα ακριβώς αυτό προσπαθούμε να ξεπεράσουμε με την λεγόμενη έξυπνη ρυθμιστική ατζέντα. Εδώ για να δείτε μια εικόνα του τι μπορεί να γίνει για να μειωθούν οι φραγμοί. Αλλά βεβαίω θα πρέπει να δούμε και το διοικητικό κόστος. Το κόστος όμως δεν μπορούμε να το δούμε μεμονωμένο, γιατί πρέπει να δούμε και το τι κάνουν οι πράξεις μας. Γιατί αυτό το οποίο ενδιαφέρει τελικά τις επιχειρήσεις μπορεί να μην είναι μόνο το κόστος, αλλά η ευκολία στο να λειτουργήσουν. Και βέβαια αυτό τελικά επιδρά και τη δημόσια διοίκηση και τους πολίτες ως φορολογούμενους. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό το οποίο ονομάζουμε έξυπνη ρύθμιση. Ε, συχνά μετράμε το κόστος και το όφελος και το όφελος θα πρέπει να υπερβαίνει το κόστος και με μια στρατηγική στόχευση μπορεί να γίνει αυτό. Πρέπει λοιπόν να ε, ορίζουμε σωστά τις ε, προτεραιότητές μας και αυτό ακριβώς προσπαθεί να μας δείξει το διάγραμμα. Υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες οι οποίες θεωρούμε ότι μπορούν να μετρήσουν αντικειμενικά το όφελος κάποιων κανονισμών, αλλά ίσως να μην συμπίπτουν πλήρως με τις υφιστάμενες δραστηριότητες που υπάρχουν. Υπάρχουν πράγματα που θα έπρεπε να γίνουν ε, και θα έπρεπε να σταματήσουν και ε, πράγματα που γίνονται και δεν ευθυγραμμίζονται με τις ε, δραστηριότητες. Το κόστος λοιπόν των επιχειρήσεων θα έλεγα πως ξεκινάει από κάτω προς τα πάνω. Υπάρχει ένα τυποποιημένο μοντέλο κόστους που μετρά το τι κοστίζει η ρύθμιση στον κάθε κλάδο θα έλεγα είναι μεγάλες οι διαφορές ανά ναι. κλάδο βλέπουμε τον χρηματοπιστωτικό, τον φαρμακευτικό, την γεωργία δεν μπορούμε όμως να διακρίνουμε μεταξύ φραγμών που είναι απαραίτητοι ε, βάρη θα έλεγα που είναι απαραίτητα για να επιτύχουμε μια μείωση των φραγμών και βάρη τα οποία ε, δεν χρειάζονται και μπορούν να καταργηθούν. Στη δεύτερη στήλη βλέπετε όμως πως υπάρχει μια δυνατότητα μείωσης ε, αρκετά μεγάλη. Έχουμε, ε, εδώ πέρα το έχουμε ονομάσει βεβαίως μείωση που έχουμε επιτύχει. Ήταν η μείωση που θα μπορούσαμε να επιτύχουμε αν τα κάναμε όλα αυτά. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να δούμε το κόστος και τους φραγμούς. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη ναι. ε, εδώ παραβαστήκαμε σε μία έρευνα, καταλήξαμε στους 10 ε, πιο επιβαρυντικούς ε, κανονισμούς που συχνά συμπίπτουν με αυτούς που έχουν τους περισσότερους φράγμους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βλέπουμε εδώ πέρα πως ε, έχουν διαφορετικές προτεραιότητες, ίσως να μην είναι τόσο παρούσες στους ε, τομείς αυτούς, αλλά δεν μπορούμε, όπως είπα, να διακρίνουμε μεταξύ των απαραίτητων βαρών και άλλων που θα μπορούσαν να περικοπούν δραστικά. Οπότε αυτό είναι ένα αναλυτικό βήμα που πρέπει να γίνει. Συνοψίζοντας. Τι ξέρουμε, εντάξει, μπορεί να μειωθεί το κόστος και ξέρουμε από τις διεθνείς συγκρίσεις πως ε, υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκές χώρες. Κάποια κράτη-μέλη τα πάνε καλά. Υπάρχει ο δείκτης ε, της ευκολίας ε, του επιχειρήν. Διοικητικές διαδικασίες οπωσδήποτε μπορούν να απλοποιηθούν, αυτό αναγνωρίζεται, αλλά δεν έχει απαντηθεί το πόσο μπορεί ακριβώς να γίνει, μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η μείωση, γιατί πρέπει να βρεθεί η ισορροπία, όπως είπαμε, μεταξύ της απαραίτητης ρύθμισης και της περιτής. Ένα άλλο θέμα είναι η λεγόμενη προσέγγιση του κόστους της μη Ευρώπης. Το βλέπουμε δηλαδή από πάνω το τι προσφέρει η ενιαία αγορά και έχουμε εδώ πέρα ξεκάθαρες προτεραιότητες όπως την ψηφιακή εσωτερική αγορά της οποίας το όφελος υπολογίστηκε σε 450 δισεκατομμύρια ευρώ το έτος ως μια ενιαία περιοχή υπηρεσιών, αγαθών και ενιαίων ρυθμίσεων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ μεγάλες οι διαφορές βλέπετε. Μετά. Μετά. Βλέπουμε πως υπάρχουν πολλές ε, δραστηριότητες. Αυτή τα πράγματα δεν είναι καινούργια. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ποιοι είναι οι τομεί προτεραιότητας και η Κομισιόν ε, λαμβάνει δράση σε όλους αυτούς τους τομείς. Όμως, η σχέση μεταξύ δραστηριότητας και αποτελέσματος ε, συχνά δεν είναι σαφής. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο κενό που δείχνει ακριβώς ε, το... τον χρόνο που χρειάζεται η νομοθετική διαδικασία και ε, πέρα από τη διαδικασία σύνταξης υπάρχει και η διαδικασία εφαρμογής μέχρι να αρχίσει να επηρεάζει τη λειτουργία της αγοράς. Δηλαδή από την αρχή μέχρι την εφαρμογή είναι πολύ ο χρόνος. Μιλάμε για αρκετά χρόνια βλέπετε στον πίνακα και θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες δράσεις οι οποίες δεν θα είναι νομοθετικές προτάσεις. Παράδειγμα, η στρατηγική της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Αν δούμε το κόστος της μη Ευρώπης ε, όπως έχει οριστεί το κενό που υπάρχει στην ε, εσωτερική ψηφιακή αγορά. από την σχετική έκθεση από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουμε ένα κόστος 277 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι στιγμής. Αν δούμε το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ε, ενιαίας αγοράς μιλάμε ότι για ένα κόστος της ε, καθυστέρησης που θα είναι 1,5 τρισεκατομμύριο τα επόμενα πέντε χρόνια. Και η στρατηγική αυτή δεν είναι και πολύ καινούρια. Είναι συνέχεια της ψηφιακής ατζέντας για την Ευρώπη που ήταν επιτάπτωση ήδη το 2010. Οπότε έχουν γίνει πολλά πράγματα εντωμεταξύ και το κόστος ε, συνεχίζει να υφίσταται. Ένα άλλο θέμα είναι η τελωνιακή μεταρρύθμιση. Εδώ έχει υπολογιστεί το βάρος στα 87 δισεκατομμύρια και πάλι η διαδικασία αυτή τραβάει. Υπάρχει ο τελωνιακός ε, κώδικας ε, που θα εφαρμοστεί από του χρόνου αλλά η υποδομή ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος επιχειρήσεις θα ξεκινήσει από του χρόνου. Αν δούμε λοιπόν τη μελέτη αντικτύπου που είχε γίνει το 2012 κομμάτι αυτής της ε, πολιτικής βλέπουμε πως θα εφαρμοστεί το 2017 οπότε αν το πάρουμε όντως ε, της μετρητής έχουμε ένα κόστος μέχρι στιγμής ήδη 260 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένα τρίτο παράδειγμα είναι η μεταρρυνήση του ΦΠΑ. Και εδώ παρόμοια τα πράγματα. Υπάρχει πολιτική που χαράζεται εδώ και χρόνια και το κόστος συσσωρεύεται και βλέπουμε εδώ πέρα το τι γίνεται. Οι μελέτες που έχουν δημοσιευτεί λοιπόν ορίζουν κάποιες ημερομηνίε, αλλά μετά στην πράξη καθυστερούν όλα αυτά. Και μετά βεβαίως κοιτάμε τους βασικούς τομείς που σχετίζονται με την ενιαία αγορά και βλέπουμε πως πράγματι υπάρχουν δραστηριότητε και ωφέλη αλλά συχνά βλέπουμε και σημαντικές καθυστερήσεις και κενά. Και με δεδομένο το υψηλό κόστος της μη Ευρώπης όλα αυτά συσσωρεύονται σύν το χρόνο. Ε, όλα αυτά δεν θα σας τα πω τώρα εις βάθος. Λοιπόν, ε, και βέβαια υπάρχει και το θέμα της μεταφοράς ε, στο εθνικό δίκαιο. Υπάρχει το θέμα του επίπεδου εφαρμογής, δηλαδή και να περάσει η νομοθεσία. Ε, υπάρχουν άλλα προβλήματα μετά. Διαφορές στην εφαρμογή που μπορεί να είναι εξίσου βλαπτικές με τους φραγμούς. Ένα άλλο παράδειγμα. Αυτό το είδαμε στην έκθεση για την ψηφιακή στρατηγική. Το χρονοδιάγραμμα εκεί πέρα. Μάλιστα. Όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, το κόστος της μη Ευρώπης είναι 204 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο και υπάρχουν ε, νομοθετικές προτάσεις ε, και νομοθεσία αλλά υπάρχει και κάποια ορολογία η οποία είναι ασαφής σε όλες αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές ε, και τα σχετικά και δεν ξέρουμε πώς θα χρειαστεί για να καρποφορήσουν όλα αυτά. Αν είναι λοιπόν να το πάρουμε σοβαρά αυτά, το κόστος της καθυστέρησης είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως έχουν σημασία οι ποσοτικοποιημένες μελέτες ε, αντικτύπου για να έχουμε προτεραιότητες, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Και βεβαίως ε, το να υπολογίζουμε το κόστος ε, της αδράνειας είναι κάπως δύσκολο γιατί και τα στοιχεία βρίσκονται σε διάφορες εκθέσεις, ε, διάβλους και πηγές. Επίσης πρέπει να γίνεται και μια αξιολόγηση εκ των υστέρων. Για να δούμε δηλαδή αν λαμβάνονται οι δράσεις ε, στους κατάλληλους κλάδους, αν είναι σωστές οι προτεραιότητες. Ε, σας έδειξα πριν το διάγραμμα, μπορεί να υπάρχει ένα κενό πολιτικής να γίνεται λανθασμένη κατανομή των πόρων. Αυτά πρέπει να αξιολογούνται ξανά και ξανά. Και τέλος βεβαίω το κόστος καθυστέρησης, ε, της καθυστέρησης είναι πάρα πολύ ψηλό. Και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου και να διαμορφώσουμε ανάλογα την χάραξη της πολιτικής. Υπεραιτέρω τώρα μείωση του κόστους ε, και των φραγμών. Ναι. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε κάποιου τομείς προτεραιότητας για να χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά τον χρόνο σας. Αλλά πρέπει να αντιληφθούμε καλύτερα και το πού πρέπει να εστιάσει η δράση. Δηλαδή, σημαντική η φραγμή της αγοράς, αλλά πρέπει να γίνουν πιο κατανοητοί. σαφώς ε, η ρυθμιστική φραγμή ε, συχνά είναι ξεκάθαροι στόχοι. Υπάρχουν ε, διάφορες δράσεις που μπορούν να γίνουν. Και υπάρχει σχεδόν πλήρης συνένεση για το τι μπορεί να γίνει. για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παραδείγματο χάρη, οι νόμοι για τις πωλήσει κτλ. Ένα άλλο στοιχείο σημαντικό είναι ο ρόλος της ε, πληροφορικής και της τεχνολογίας επικοινωνιών. Τα δίκτυα δηλαδή, αλλά και η ανάλυση πέρα από τη δικτύωση. Και ο ρόλος της τεχνολογίας αυτής είναι διτός. Γίνεται πιο αποτελεσματική η διαδικασία χάραξης πολιτικής μέσω της ορθής κατανομής πόρων αλλά και άμεσα μέσω της μείωσης του κόστους και αποτελεσματικότητας της διοίκησης μετά υπάρχουν πολλά εργαλεία ηλεκτρονικής ε, διακυβέρνησης εμείς θεωρούμε πως ε, μπορεί να γίνει καλύτερη χρήση των εργαλείων αυτών ε, έτσι ώστε πραγματικά να μπορέσουν να οθήσουν τον κύκλο χάραξης πολιτικής αλλά να έχουμε και μια διαρκή ενημέρωση για την ύπαρξη φραγμών και την εμφάνιση νέων και έχουμε κάποιες συστάσεις εδώ. Ναι, ναι. Πολλά από αυτά τα δεδομένα δημιουργούνται από τις ε, συμβουλές μας δίνει το Enterprise Europe και LP. Μας ζητήθηκε συγκεκριμένα να κοιτάξουμε τον ρόλο της διαδικασίας ε, της διαβούλευσης. Και θεωρούμε πως ε, συγκεκριμένες προτάσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν γρήγορα όπως και κάποια ζητήματα ουσίας κάτι το οποίο δεν είναι σαφές ακόμα και θα έπρεπε να υπάρχει μια υποχρέωση ε, αλλαγές στην ομοθεσία να είναι όρατες και να συνδέονται και με τα εφαρμοστικά μέτρα ή με τα Υπάρχουν και κάποια άλλα πρακτικά ζητήματα σε σχέση με την διαβούλευση. Θεωρούμε πως πολλά πράγματα μπορούν να βελτιωθούν στην εφαρμογή. ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους πολίτες, ε, μη μονομένους πολίτες. Λοιπόν, και πάλι βλέπουμε πως η ανάλυση των πληροφοριών που συλλέγονται είναι πάρα πολύ σημαντική και υπάρχει, όπως είπα, η δυνατότητα τέτοια προχωρημένων αναλύσεων. Λοιπόν, εδώ έχουμε την πλευρά της χάραξης πολιτικής. Αν δούμε τώρα το κόστος, το άμεσο αντίκτυπο της τεχνολογίας πληροφορικής στη του κόστους, είδαμε κάποια παραδείγματα. Την Εστονία, την Κορέα. Ε, ένα παραδείγμα, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες στις οποίες ε, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι προχωρημένη στην Ευρώπη. Απλά μας δίνει κάποια παραδείγματα του πώς η έξυπνη χρήση της τεχνολογίας πληροφορικής μπορεί να μειώσει το διοικητικό άχθος στις επιχειρήσεις άλλη περιπλοκή που βρίσκουμε είναι πως ε, οι πρωτοβουλίες στο εθνικό επίπεδο έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν νέους φραγμούς. Δηλαδή να δημιουργήσουμε υποδομές σε μία χώρα που μπορεί να ωφελήσουν τις επιχειρήσεις ε, σε αυτή τη χώρα μπορεί αυτό να είναι ένα σφραγμό στην ολοκλήρωση της αγοράς. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός στο ευρωπαϊκό επίπεδο και μια διαλειτουργικότητα. Οπότε υπάρχει μια ευρωπαϊκή ευθύνη εδώ. Τι θα λέγαμε λοιπόν το κόστος της ε, καθυστέρησης ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν το έχουμε δώσει την προσοχή που αξίζει και είναι ουσιαστικό. Οπότε εμείς θα λέγαμε πρώτα απ' όλα να υπάρξει μεγαλύτερη ε, ορατότητα θα έλεγα αυτού του πράγματος γιατί βεβαίως το κόστος της μη Ευρώπης είναι σημαντικό αλλά το κόστος της καθυστέρησης σημαίνει πως η δράση πρέπει να αναλυφθεί γρήγορα και πραγματικά ξαναρίχνει το βάρος στην διαδικασία χάραξης πολιτικής. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αποφασιστεί να αναλυφθεί η δράση, αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα. Και βέβαια το κόστος της ε, καθυστέρησης είναι ότι πρέπει να καλύψουμε όλους τους τομείς ε, δράσης και να υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και αυτό μαζί με την στρατηγική διαδικασία χάραξης προτεραιοτήτων είναι οπωσδήποτε ένας, είναι ένα μεγάλο όφελος για την ευρωπαϊκή οικονομία. Και κάτι που σχετίζεται με αυτό. Έχουμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το κόστος ε, της ε, τεχνολογίας ε, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και έναν διτό ρόλο, δηλαδή τη χάραξη προτεραιοτήτων και μια στρατηγική ευθυγράμμιση και βεβαίως άμεση και απευθείας μείωση του κόστους και των φραγμών. Και θεωρούμε ότι όπως είδαμε πριν υπάρχει δυνατότητα μείωσης του κόστους και σε κάποιες περιπτώσεις ε, το διοικητικό κόστος ε, μπορεί να είναι μηδέν για κάποιους ε, στόχους πολιτικής. Θεωρούμε λοιπόν πως εδώ πέρα υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών. Αρκεί να είμαστε τολμηροί, γιατί όπως είδαμε στην Εσθονία αν κάποιος ε, ζητάει φοιτητικό δάνειο τα στοιχεία προσυμπληρώνονται με βάση την διαθεσιμότητα του δικτύου από διάφορες πηγές του κράτους και προσυμπληρώνονται επίσης οι φορολογικές δηλώσεις ε, κατά το οποίο μπορεί να ωφελήσει πάρα πολύ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ειδικά για τον ΦΠΑ και τη συμμόρφωση την τελωνιακή. γιατί ακριβώς πολλά από αυτά τα πράγματα ε, βρίσκονται ήδη επιτάπητος και μπορούν να ελαφρύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καλά. Ε, υπάρχουν ερωτήσεις? Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που ετοίμασαν την ε, έκθεση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. και μας φέρνει ενώπιον μια σκληρή πραγματικότητα και γι' αυτό θα συνεχίσω στα Ολλανδικά. Βλέπουμε εδώ πέρα πως πραγματικά το μήκος, το χρόνος που απαιτείται μέχρι να νομοθετήσουμε είναι πάρα πολύ ε, μεγάλος. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι το κόστος καθυστέρησης είναι τεράστια νούμερα, 240 δισεκατομμύρια το χρόνο. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε βάρος στην ψηφιακή εσωτερική αγορά, γιατί βλέπουμε πως ε, πρέπει και η νομοθεσία να είναι future proof. Και βεβαίως δεδομένου του πόσο γρήγορα αλλάζει ο κόσμος της ε, τεχνολογίας ε, μάλλον αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να προσαρμοστούμε και να νομοθετούμε γρηγορότερα και οι διαδικασίες του Κοινοβουλίου επίσης πρέπει να γίνουν πιο γρήγορες θεωρώ πως τα νούμερα αυτά μιλάνε από μόνα τους Ακούσαμε επίσης ε, τα της διοργανικής ε, συμφωνίας που συμφωνήθηκε προχτές. Δεν ξέρω όμως αν πάει στη σωστή κατεύθυνση. Είδαμε εδώ πέρα πως ε, είναι πάρα πολύ σημαντική η διαδικασία της διαβούλευσης που επίσης είναι αργοκίνητη. Δεν υπάρχει νομίζω επίσης ε, αρκετή καινοτομία. Θα μπορούσε ε, να γίνεται ηλεκτρονικός. του χάρη, δυστυχώς δεν γίνεται όμως. Πρέπει λοιπόν να αντλήσουμε τα διδάγματά μας από αυτή τη μελέτη. Να κινηθούμε γρήγορα. Και να είμαστε αποτελεσματικοί όχι μόνο λόγια και σχέδια δράσης που δεν εφαρμόζονται. Έχω τώρα και δύο συγκεκριμένες ε, ερωτήσεις για την καλύτερη νομοθεσία. Θα ήθελα να ρωτήσω τους συντάκτες της μελέτης για το εάν ένα σαφής για τη μείωση του διοικητικού άχθους εσείς μιλήσετε παραδείγματο χάρη για το 25% ε, θα ήταν κάπου σε αυτό το ύψος και η δεύτερη ερώτηση για τον ΦΠΑ Αντιλαμβάνω πως είναι δύσκολο το ότι υπάρχουν διαφορετικά συστήματα ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο και θα πρέπει να πάμε σε κάποια αναρμόνιση των συστημάτων των κρατών μελών. Αλλά πριν από αυτό θα υπάρξει ένας συντονισμός. Και το ερώτημά μου είναι... κάτω την άποψή σας μπορεί να υπάρχει παραδείγματος χάρη ένα one-stop shop που θα ορίζεται ο ΦΠΑ θα βοηθούσε κάτι τέτοιο. Ο Νίκολα. Ναι, θέλω να κάνω τις εξής ε, σκέψεις. Πρώτα απ' όλα, ότι κάθε φορά που παρουσιάζονται μελέτες αυξάνεται όλο και το κόστος της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ψυχολογικό, ε, μάλλον της μη Ευρώπης. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ψυχολογική πίεση για να κάνουμε περισσότερες νομοθετικές ρυθμίσεις. Από την άλλη είμαστε εμείς συνομοθέτες στην Ευρώπη και θα πρέπει την ίδια μελέτη να την δει, βλέπουν και τα κράτη-μέλη να αντιληφθούν και οι κυβερνήσεις ότι το κόστος ε, της Ευρώπης ε, ή της μη Ευρώπης εξαρτάται όχι μόνο από το Κοινοβούλιο αλλά και από το Συμβούλιο. Ένα θέμα δεν συζητούμε επαρκώς και το ανέφερε η προραλήσασα και βλέπω ότι εάν δεν συζητήσουμε το θέμα της φορολογικής εναρμόνισης μια και στην Ευρώπη υπάρχουν χώρες οι οποίες πράττουν ε, και θα χρησιμοποιήσω μια σκληρή έκφραση φορολογικό dumping, συγχωρήστε μου την ε, έκφραση και από την άλλη υπάρχει προσπάθεια μέσω φραγμών και εμποδίων να εμποδίσουμε την ε, είσοδο εκείνων που έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω της πιο ευεργετικής φορολογικής νομοθεσίας δεν νομίζω ότι προχωρούμε προς μια εσωτερική αγορά και προς μια Ευρώπη πιο ολοκληρωμένη. Εδώ έχουμε ένα, να κάνουμε έναν στόχο τον οποίο θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με τη, με τη φορολογική εναρμόνιση. Σάλτε Μόζερ. Πρόεδρε, ήταν όντως πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση της μελέτης. Αλλά δεν μας δίδαξε και τίποτα το καινούριο. Τα ίδια ακούμε εδώ και χρόνια. Βασικό συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει εύκολη λύση. Κρατάει πολύ καιρό όλη αυτή η ιστορία. Πρέπει να κάνει προτάσεις η Επιτροπή, όταν κατατίθενται αυτές δεν είναι αρκετά συγκεκριμένες. Καιρό τώρα βλέπουμε ότι ε, οι διαδικασίες από την ώρα που εντοπίζεται ένα πρόβλημα μέχρι την ώρα της ανάληψης δράσης είναι υπερβολικά μακροχρόνιες. Χρειάζεται λοιπόν πιο γρήγορη δράση. Οι καθυστερήσεις, ναι, τις αναφέρατε κι εσείς και θα συμφωνήσω. Ταυτόχρονα είναι πιστεύω δύσκολο να διαγνώσει κανείς τι πρέπει να συμβεί για να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Έχουμε πάνω από 500 εκατομμύρια πολίτες, πάνω από 700 βουλευτές, πάνω από, έχουμε 28 κράτη-μέλη. Ε, κάπως πρέπει να συνοηθούν όλοι αυτοί. Και φτάνουμε έτσι στο ερώτημα. Θα πρέπει βεβαίως πάντα να προσπαθούμε να βελτιώνουμε τις διαδικασίες και όλα αυτά. Αλλά, αλλά δεν είναι δυνατό να πατάμε ένα κουμπί και να ε, προχωράει κατά τρόπο αυτοματοποιημένο και απρόσκοπτο η νομοθεσία, γιατί πάλι, πάλι κάπου υπάρχει ένα καινούριο στοιχείο. Και ένα παράδειγμα, η Ισλανδία. Με ένα καταπληκτικό επίπεδο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η Εσθονία. Η Εστονία που έχει ένα πολύ καλό επίπεδο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με κανόνες που λειτουργούν πολύ καλά για την ίδια την εστονική αγορά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι άλλες επιχειρήσεις εκτός Ισλανδία, ε, Εστονίας μπορούν να ε, έχουν την ίδια ε, εύκολη πρόσβαση. Αντιθέτως μπορεί να υπάρχουν εμπόδια, μπορεί να υπάρχουν φραγμοί. Αυτούς πρέπει να τους καταργήσουμε. Και ίσως μια λύση ήταν να προτείνουν τα κράτη-μέλη ε, ε κίνητρα με κάποια ιδέα αμοιβαιότητας, ώστε να βελτιώνεται η κατάσταση και να απαλήφονται οι φραγμοί μεταξύ τους. Ξέρουμε πολύ καλά ότι για τα εμπόδια αυτά στην εσωτερική αγορά υπεύθυνο είναι επιτοπλίστων το Συμβούλιο. Εκείνο, το, εκείνο είναι το οποίο δεν διευκολύνει την κατάσταση. Άρα θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες στην αγορά και την ταχύτερη βέβαια έγκριση νομοθεσίας. Μα Χρήστα, μόλις έχασες μια σημαντική παρουσίαση από την Κομισιόν για τις παραβιάσεις και ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν προηγουμένως ήταν να διασφαλίζουμε ότι είναι σωστή η νομοθεσία μας από την αρχή. Για να μπορεί καταρχάς να εφαρμοστεί, να είναι εφαρμόσιμη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Κρίμα που την έχασες ρε παιδί μου. Συγγνώμη που διέκοψα, αλλά Ορίστε λίγο καλύτερα. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι πολύ πολύ πλοκό θέμα. Πολύ πλοκό. Το συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι απολύτως απαραίτητο να παίρνουμε πάντα, κάνουμε πάντοτε τα σωστά βήματα για να ωφελούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όλοι οι εταίροι η ψηφιακή στρατηγική για την εσωτερική και η στρατηγική της εσωτερικής αγοράς πρέπει να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Εκτιμώ ιδιαίτερα αυτές τις αναλύσεις και θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτή την υψηλής ποιότητος παρουσίαση. Ήταν πολύ καλή η έμφαση που δόθηκε για το πρόβλημα ακριβώς αλλά όπως είπε και ο συνάδελφός μας Δάντης η σωστή νομοθεσία θα έλυνε τα προβλήματα και δεν υπάρχει αυτό αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι τρέχουμε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει. Λένε να λύνουμε πρώτα τα προβλήματα και μετά να αρχίζουμε να παίρνουμε μέτρα. Εδώ προτρέχουμε πολύ, προτρέχουμε. Ακούσαμε για μεθοδολογία, ακούσαμε πώς θα μπορούσαν να βοηθηθούν όσοι πλήττονται από αυτά, πόσοι θα μπορούσαν να βοηθηθούν από τη συμπλήρωση του φορολογικού των δελτίου και σε διαμεθοριακές περιπτώσεις και υπάρχουν και, άλλα, και άλλες περιπτώσεις όπου θα μπορούσαμε να είχαμε μικρές επιτυχίες. Χρειαζόμαστε ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και διορίες. Καλό θα ήταν επίσης τα προβλήματα αυτά να τα βλέπουμε τομέα τον τομέα. Όλους τους τομείς για να δούμε ποια είναι τα προβλήματα και άρα και ποια είναι τα καταλληλότερα μέτρα. Ακούσαμε επίσης πώς θα μπορούσαμε να διαλύσουμε, να διορθώσουμε, να αφαιρέσουμε τους φραγμούς που υπάρχουν και ότι ό,τι κόστος χρειαστεί για τις καθυστερήσεις είναι δικαιολογημένο. Θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντική είναι η τομεακή προσέγγιση. Ας πούμε η φαρμακοβιομηχανία είναι βιομηχανία που απαιτεί πάρα πολλούς πόρους, είναι ποροφόρα. αλλά υπάρχει και μεγάλη συγκέντρωση σε αυτήν και αυτό θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα για την έρευνα για αυτές τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν δύσκολη κατάσταση. Βέβαια υπάρχουν ευρεσιτεχνίες αλλά, και προστατεύονται αυτές, αλλά όχι αρκετό χρόνο ώστε να έχουν κέρδος, το κέρδος που πρέπει. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η στρατηγική να συμπεριλαμβάνει πρόσθετα πιστοποιητικά και ε, διπλώματα ευρεσιτεχνίας που να επιμικίνουν το χρόνο της προστασίας. Επίσης πρέπει όλα αυτά να εναρμονιστούν, να συντονιστούν, να τύχουν συντονισμού με έναν κοινό στόχο και με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και διορίες. Αυτό είναι ο μόνος τρόπος να πετύχουμε. Και οι καθυστερήσεις πρέπει να αποφεύγονται. Αυτό θα ωφελούσε όλες τις χώρες μέλη Και η διαφάνεια και η διαφάνεια. Ναι, ευχαριστώ για την παρουσίαση. Θέλω και εγώ να κάνω μερικά σχόλια. Πρώτα απ' όλα βέβαια είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε μια πολύ λεπτομερή εικόνα, μια αντικειμενική εικόνα, ως οικονομολόγος και μαθηματικός όμως, με προβληματίζει κάποια, κάπως η βάση των επιχειρημάτων σου. Βεβαίως το κόστος της απουσίας της Ευρώπης είναι χρήσιμο, να το βλέπουμε, δηλαδή αν υπάρχει κοινή δράση, πόσο πιο πολλές οικονομίες θα είχαμε. Εσύ όμως θεωρείς ότι η δράση θα ήταν σύμφωνη με τα πιθανά ωφέλη που καταγράφεις στη μελέτη. Αλλά δεν είναι δυνατό να θεωρήσουμε ως αξιωματική αρχή ότι κάθε δράση θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Λες Φερρυπίν ε, ΦΠΑ. Ε, ναι, αλλά από την εμπειρία που έχουμε και από φέτος ακόμα, ακόμα ήταν ότι πολλές μικροεπιχειρήσεις σταμάτησαν να πολλούν στην Ευρώπη με την εισαγωγή εφέτος αυτών των συστημάτων για το ΦΠΑ. Και επίσης, η Αρλή νομίζω ανέφερε, ότι ένας από τους κύριους τομείς αποδέσμευσης αξίας θα ήταν η απελευθέρωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το ανέφερε και Αρλίν. Ναι, αλλά αυτό προϋποθέτει εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του αγοραστή για την ε, διαγραμμική του αγορά. Εχθές μόλις η Επιτροπή κατέθεσε πρόταση για τα υλικά αγαθά, όπου ορίζονταν διαφορετικοί κανόνες αγοράς ενός αγαθού, τηλεφώνου και το καθεξής, διαγραμμικά ή Και βέβαια επισημάνθηκε ότι αυτό οδηγεί και σε σύγχυση και σε ε, κατακαιρματισμό και υπονομεύει την εμπιστοσύνη και ενώ είχε υποθεί ότι θα αναλυφθεί καμία δράση σε σχέση με την ε, εσωτερική αγορά εφέτος και ενώ έχουμε κλείσει το πακέτο για τις τηλεπικοινωνίες και ελπίζω ότι αυτό θα είναι χρήσιμο για να μπορέσει ο κόσμος να ταξιδεύει στην Ευρώπη χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Τώρα έχουμε κλείσει και το πακέτο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, δηλαδή καλύτερη αντοχή και ανθεκτικότητα σε σχέση με την κυβερνοασφάλεια αλλά ταυτόχρονα με ανησυχεί το γεγονό ότι η προστασία των δεδομένων που θα έρθει την επόμενη εβδομάδα και που έχει κέρια σημασία θα κριθεί και κλεισμένα των θυρών χωρίς να ενημερωνόμαστε όλοι εμείς που δεν θα είμαστε κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Και από την άλλη μας λέτε ότι αν κάτι δεν πάει καλά, θα έχει συντριπτικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις και δεν τις μικρομεσαίες. Άρα λοιπόν πρέπει και να είναι σωστή η διαμόρφωση διατύπωση της νομοθεσίας και να είναι τέτοια που θα αποδεσμεύσει τις δυνάμεις αγοράς και δεν θα ε, δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προβλήματα. Και πρέπει να αξιολογηθεί σωστά η συνέπεια κάθε νομοθετήματος. Αυτό λοιπόν με ενδιαφέρει, ιδιαίτερα δε αυτό που λέτε για, την εξε, για τις εξελίξεις στην Εσθονία που δείχνουν πώς μπορεί μια χώρα ε, να έχει πολύ καλές επιδόσεις και χωρίς παρέμβαση νομοθετική, γιατί έχει και αυτό πολύ μεγάλη σημασία. Θέλετε να έρθετε στο, να περάσετε σε κάποιες από τις ερωτήσεις μας. Και σας ευχαριστώ πολύ για, τις, για την παρουσίαση. Απάντηση. Ναι, όντως. Εύστοχο αυτό που υπόθηκε για το κόστος της απουσίας της Ευρώπης σε σχέση με κάποιους τομείς πολιτικής όπου δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς η δράση μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα. Πρέπει να κοιτάξουμε τις στρατηγικές που έχει αναπτύξει η Ένωση και πώς έχουν υλοποιηθεί αυτές για να προσαρμόσουμε αντίστοιχα στην εσωτερική ψηφιακή αγορά. Η προσέγγιση δηλαδή είναι η εξή. Εάν όλες οι δράσεις σε ένα τομέα πολιτικής τίνουν στην ε, κάλυψη του χάσματος ή της απουσίας της μη Ευρώπης κτλ. καταγράφεται αντίστροφα το κόστος της καθυστέρησης. Δηλαδή και οι δράσεις πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις προτεραιότητες σε ένα πρώιμο στάδιο. και για κάθε μέτρο θα πρέπει να καταγράφονται τα ωφέλη του και το κόστος από την μη εισαγωγή του ή από την απουσία Ευρώπης. ευχαριστώ πολύ, μας βοήθησε πολύ αυτό. Τώρα θα δώσω την Προεδρία στον κύριο Δάντη. Ευχαριστώ πολύ και καλά Χριστούγεννα. One more comment from the One more Yeah. Okay, thank you. Um, <coughs> uh, one of the members uh, raised the question. Ευχαριστώ. Κάποιος βουλευτής είπε κάτι για την Εσθονία. Και τα καλά, το καλό παράδειγμα της Εστονίας. Και βέβαια υπήρχε και το σχόλιο για το εάν τα κράτη-μέλη αν δρουν μόνα τους δημιουργούν φραγμούς για τα άλλα κράτη-μέλη. Είδα λίγο κάποιες οικονομίες που είχαν γίνει στην Εστονία. Και ένα από τα παραδείγματα είναι το ηλεκτρονικό μητρό επιχειρήσεων. Τώρα λοιπόν μπορούν οι επιχειρήσεις ε, να τα κάνουν όλα αυτά επιγραμμικά. Και ε, γίνεται σε 20 λεπτά η υπόθεση. Ε, μάλιστα τους έχει γράψει το βιβλίο Guinness για την εγγραφή στο Μητρό Επιχειρήσεων. Αυτό το οποίο έχει κάνει εστονική κυβέρνηση είναι ότι έχει ανοίξει αυτή τη διαδικασία σε εταιρείε από άλλα κράτη-μέλη. Οπότε εταιρείε από άλλα κράτη-μέλη ε, εγγράφονται επίσης πάρα πολύ γρήγορα και έχουν διμερείς ε, συνεννοήσεις με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε και οι εστονικές εταιρείε ε, να εγγράφονται στα άλλα κράτη-μέλη. Ναι. Κάποια παραδείγματα τώρα για το πώς μπορούμε να δούμε αυτά τα διασυνοριακά ζητήματα. Νομίζω υπόθηκε ε, δεν... Καλό είναι να μην έχουμε μια κατάσταση όπου το κάθε κράτος μέλος ή λίγα-λίγα τα κράτη-μέλη να κάνουν δικές τους ρυθμίσεις μπορεί να είναι καλές αλλά τελικά θα είναι φραγμή για τα άλλα κράτη-μέλη. Λοιπόν, ε, εμένα με συγχωρείτε πρέπει να φύγω για να συναντήσω εστονούς επιχειρηματίες. Ehm, Έχουμε λοιπόν το τελευταίο σημείο και σας ευχαριστώ για την ενημέρωση και την μελέτη. Τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ερώτηση της ε, κυρίας Κοράου, του κυρίου Κοράου. Ε, πολύ ενδιαφέρουσα. Θα του δώσω το λόγο για να μας παρουσιάσει την γραπτή του ερώτηση και μετά η Επιτροπή παρακαλώ. Κοράου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Δάντη. Και εδώ και μερικά χρόνια, λιγότερο από μια δεκαετία, η Ιταλία δεν έχει μπορέσει ακόμη να αντιμετωπίσει το ζήτημα των εκχωρήσεων των παραθαλασσίων ε, περιοχών και ακτών. Έχουμε να κάνουμε με έναν στρατηγική σημασία στο ΜΕΑ της ε, πατρίδας μας, όπου δεν ε, μπορεί να γίνει προγραμματισμός και δεν υπάρχει βεβαιότητα ως προς τις επενδύσεις. Περιμένουμε λοιπόν την έκβαση των προσφυγών που έχουν γίνει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά και από πλευρά μα προσπαθούμε να ενισχύσουμε το μέλλον του τομέα για να έχουμε μια αηφορία και καλύτερη λειτουργία. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιε είναι οι διαφορέ στην προσέγγιση σε σχέση με άλλες χώρες όπως Ισπανία, Πορτογαλία, Κροατία, σε σχέση με την κατάλληλη περιορισμένη χρονική διάρκεια αυτών των, των παραχωρήσεων χρήσης ε, που ασφαλώς ξεπερνούν τα 7, την 7 ετία που ορίζεται στην Ιταλία. Τι συμβαίνει σε σχέση με τη διαδικασία επιλογής όπου το άρθρο 12.2 της οδηγίας Μπόλκενστάιν αποτελεί μια εναλλακτική στη δημόσια προκήρυξη, στο δημόσιο Τι γίνεται σε σχέση με το άρθρο 12.3 της ε, οδηγίας Μπόλκενστάιν για την προστασία του περιβάλλοντος και της ε, πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και, της κοινωνική, και την κοινωνική πολιτική. Υπάρχουν κριτήρια προτίμησης ε, των ε, πλειοδοτών οι οποίοι θα προσέφεραν καλύτερες συνθήκες κοινωνικές κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ συνοπτική η παρουσίαση και τις ερώτησεις Η Επιτροπή ποιος θα αναλάβει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη που δεν έχουμε ακόμη ε, φτά, ε, αποστείλει γραπτή απάντηση. Ε, βεβαίως γνωρίζουμε τους κανόνες και τους σεβόμαστε και θα στείλουμε το χειρότερο δυνατό γραπτή απάντηση. Τώρα, επί της ουσίας, γίνεται λόγος εδώ για δημόσιο αγαθό, δημόσιο χώρο, δηλαδή τις ακτές, της Ιταλίας για τις οποίες δίνεται η άδεια από τις αρχές για χρήση τους για ευρωπαϊκούς στόχους. Είμαστε σε ένα διαρκή διάλογο με τις Ιταλικές αρχές. Αξιολογούμε την κατάσταση στα λοιπά κράτη-μέλη πέραν Ιταλίας και χωρίς να θέλω τώρα να προδικάσω την τελική απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για ένα κέριο ζήτημα και δι' Πρέπει να περιμένουμε τι θα πει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί εκλήθη το Δικαστήριο να απαντήσει σε δύο ερωτήματα. Πρώτον, εάν το άρθρο 2, 12 ε, της Οδηγίας περί ισχύει νέου και εάν ισχύει, προβλέπει την, ε, το παραδεκτό της αυτόματης ανανέωσης των σχετικών εκχωρήσεων δυνάμει του άρθρου 12 ε, η οδηγία περί ναι. Περιμένουμε λοιπόν την απάντηση του δικαστήριου του Λουξεμβούργου και από εκεί και πέρα θα αναλάβουμε δράση αναλόγω. Τώρα, οι υποθέσει είναι 158, C158. Ε, προδικαστικό ερώτημα από τους Ιταλούς δικαστές προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έγινε η ακρόαση της 3 Δεκεμβρίου με πολλά ερωτήματα επί της ουσίας και αναμένονται ε, συμπεράσματα από τον εισαγγελέα, προτάσει του εισαγγελέα στα τέλη Φεβρουαρίου. Αυτό είναι το κύριο σημείο για μας. Αυτά, αυτά θα κρίνουν την υπόθεση δηλαδή για μας. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλες γραπτές ερωτήσεις στις οποίες έχουμε ήδη απαντήσει. Μην να μένει λοιπόν κανείς ότι πρόκειται να αλλάξουμε γραμμή. Αλλά υπογραμμίζω ότι αυτή τη στιγμή την μπάλα την έχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου και από εκεί θα λάβουμε τις ε, ε, υποδείξεις και τις ενδείξεις για το προς τα που θα πρέπει να κινηθούμε. Εν τω μεταξύ ελπίζουμε ότι και οι ιταλικέ αρχές θα είναι σε θέση από μόνες τους να βρουν μια σωστή λύση. Καλά. ρωτάω αν θέλει κανείς το λόγο για την απάντηση που δόθηκε τώρα. Ουχή, εκ των παρισταμένων. Ας λάβει λοιπόν ο κύριος Κοράου το λόγο. Αν ε, μου επιτρέπει μάλιστα θα ήθελα και εγώ να προσθέσω κάτι όταν ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, δεν μπορώ να πω ότι είμαι και ικανοποιημένος από την πρόταση της Επιτροπής. Ασφαλώς και πρέπει να περιμένουμε την απόφαση, την προδικαστική κρίση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά και η Επιτροπή έχει ένα ρόλο αρκετά ξεκάθαρο δραματίσει εδώ. Έχουμε ένα συγκεκριμένο ερώτημα υποβάλει, πρέπει να λάβουμε και συγκεκριμένη απάντηση το Κοινοβούλιο στη τελευταία ανάλυση ε, ασκεί ελεγκτική δραστηριότητα και δίνει και τα κίνητρα προς την Επιτροπή για να αναλάβει και εκείνη από πλευρά τη δράση. Ε, άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνουμε ένα τέτοιο φαινόμενο και όχι μόνο στη δική μας Επιτροπή, αλλά και σε όλες τις Επιτροπές βλέπουμε να αντιμετωπίζουμε προβλήματα τέτοια από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με το δυναμικό των ανθρώπων που έχει η Επιτροπή στη διάθεσή της, δεν είναι παραδεκτό να μας, κάνετε, να μας δίνετε τις απαντήσεις. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Κοράου. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τη δυσθυμία μου, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα στην Ιταλία και το λέω προς τους συναδέλφους είναι ένα θέμα το οποίο συστιάται πάρα πολύ μπορεί να υπάρχουν και πολύ καλοί λόγοι για τους οποίους ε, δεν θέλει να παρέμβει στο θέμα αυτό η Ευρώπη αλλά είναι απαραίτητο το γεγονός ότι προβλέπονται εξαιρέσει ω προς την υλοποίηση την εφαρμογή αυτής της οδηγίας για 20, 30, 40 και βάλε περιπτώσεις και γι' αυτό θα έπρεπε η Επιτροπή να μας έχει δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Υπάρχουν παρεκκλήσεις για τόσα πολλά χρόνια, παρεκκλήσεις που ξεπεράνε και τα 50 χρόνια για ορισμένα κράτη και ορισμένους τομείς σε σχέση με την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Θα θέλαμε πολύ πιο συγκεκριμένε απαντήσεις, διότι η διαχείριση του θέματος αυτού στην Ιταλία είναι άκρους περίπλοκη και διοικητικά και διαδικαστικά σε σχέση με τις ίδιες τις προκήρυξεις. Και γι' αυτό, και θέλω να το πω και νωρίτερα, σε μια άλλη συζήτηση, ότι θα πρέπει να αποτρέπουμε την ανάπτυξη προστατευτικών συστημάτων σε κράτη τα οποία έχουν καταφέρει να εγγυηθούν καλές συνθήκες απασχόλησης για πολλά χρόνια και το λέω και προς την Επιτροπή έκανε, γιατί δεν ήσασταν εδώ πιο νωρίς, έκανε η, Επιτρο... η η Τοσκάνη συγκεκριμένα έναν διαγωνισμό για την κάλυψη σε ανάγκες δημοσίων μεταφορών, αστικών μεταφορών την προκήρυξή της, μια προκήρυξη την οποία κέρδισε μια γαλλική επιχείρηση ε, που εξυπηρετεί και τον ε, Μητροπολιτικό Δήμο των Παρισίων η οποία έχει αναλάβει αυτά τα καθήκοντα, αυτή την, αυτόν τον διαγωνισμό χωρίς καν να γίνει διαγωνισμός, έχει γίνει απευθείας ανάθεση. Ε, λοιπόν, προφανώς δεν είναι οι ίδιες συνθήκες απασχόλησης ή ε, χορήγησης της, ε, ε, της συμβάσεως. Πρέπει να υπάρχουν πιο υγιείς συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ένα θέμα αυτό το οποίο δεν εξαντλείται εδώ. Θα το ξανασυστήσουμε εξάπαντος. Χαίρομαι ιδιαίτερως για την ε, παρουσίαση και την παρουσία σας εδώ και αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο μπορούμε νομίζω να κηρύξουμε το πέρα στη συνεδρίασης. Την επόμενη εβδομάδα είμαστε στο Στρασβούργο και μια και ως Επιτροπή δεν ξαναβλεπόμαστε πριν τα Χριστούγεννα. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, όπως είπε και η Πρόεδρος, το επόμενο, η επόμενη συνεδρίαση μετά την χρονιά.